Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στην Ολομέλεια για τη δημοκρατική νομιμοποίηση των ε, προγράμματων οικονομικής προσαρμογής. Να καλωσορίσω τον κύριο Λάμερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Bundestag, τον, κύριος, ε, τον κύριο Χάν, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινή ε, Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου και να καλωσορίσω και τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον κύριο Ότμαν Κάρας και τον Λουν Χουαν ε, Νόγκ, οι οποίοι όπως γνωρίζετε είναι οι συνεισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση πρωτοβουλίας για την αξιολόγηση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω συντομία ότι υπάρχουν κάρτες ε, ομιλίας ε, στα έδρανά σας, με τις οποίες μπορείτε να μας υποδείξετε ότι θέλετε να λάβετε το λόγο και ε, εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ε, κάρτα, θα πρέπει να τη συμπληρώσετε και να τη δώσετε στους κλητήρες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι με χθε το απόγευμα, δηλαδή θα δώσουμε το λόγο σε τέσσερις βουλευτές εθνικούς και στη συνέχεια θα λάβει το λόγο ένας ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως λοιπόν και να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο και συνεισηγητή της έκθεσης πρωτοβουλίας της έκθεση ε, για την ε, δραστηριότητα της Τρόικα, τον κύριο Ότμαν Κάρας, για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ε, Κύριε Αποδηματά, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι ευγνώμων που και σε αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να σας μιλήσουμε για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εξέταση ε, του ρόλου και των ε, δραστηριοτήτων της Τρόικα και ενδεχομένως να διασκεδάσουμε κάποιες παρεξηγήσεις, διότι είχα τις τελευταίες μέρες την εντύπωση ότι μας ρωτάνε «Μα επιτρέπετε, ε, να γίνεται αυτό. Ναι, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει κάθε απόφαση των θεσμικών οργάνων ακόμα και αν δεν γίνεται με βάση το κοινοτικό δίκαιο, το Κοινοβούλιο μπορεί να ελέγχει, να αξιολογεί και να βγάζει συμπεράσματα για τις μελλοντικές εργασίες. Λυπάμαι που σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης δίδεται η εντύπωση ότι η άσκηση του δημοκρατικού ελέγχου από το Κοινοβούλιο και η εξέταση του πώς, μπορεί, μπορούν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στο μέλλον θεωρούνται, ε, ε, θεωρούνται κριτικοί κατά ατόμων και θεσμικών οργάνων. Το ένα είναι μια δημοκρατική υποχρέωση και το άλλο είναι μια κρίση. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μπαρόζο είπε χθε ότι είναι σημαντικό στην συζήτηση αυτή να συζητάμε από πού ερχόμαστε. Και θα ήθελα να σας θυμίσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε πολιτικά ούτε διαφορετικά θεσμικά και οικονομικά δεν ήταν προετοιμασμένοι για μια κρίση τέτοιου μεγέθους. Κανένα οικονομικό μοντέλο δεν ήταν προετοιμασμένο για μια κρίση τέτοιες εμβέλειας. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε ότι με το Μάστριχ το 1993 και την εισαγωγή του ευρώ μείναμε στα μισά του δρόμου και την νομισματική ένωση δεν την κάναμε πολιτική, οικονομική και κοινωνική ένωση. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια κράτη-μέλη ιδιαίτερα ισχύει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, δεν τηρήθηκε και η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή δεν εφαρμόστηκε. Και χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Μπαρόζο επισήμανε ότι έπρεπε να επισκευάσουμε το σκάφος εν μέσω της θύελας. Έχουμε κάνει πολύ δρόμο, αλλά τονίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο μας. Η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή των όσων μάθαμε από την κρίση. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Τρισέ, Σε μία από τις πέντε ακροάσεις που είχε κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα είπε ότι έχουμε την μεγαλύτερη κρίση ε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς να έχουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και εάν δεν αξιολογήσουμε την Τρόικα, μάλλον χωρίς την Τρόικα θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερη κρίση όπως είδαμε στη δεκαετία του 30 ε, του προηγούμενου αιώνα. Πολλά κράτη δεν ε, έλαβαν λαμβάνουν χρήματα από τις χρηματαγορές. Πολλά κράτη δεν είναι σε θέση να καλύψουν ε, τις δαπάνες ε, της εκπαίδευσης, ε, τη υγείας, της καινοτομίας, των επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για να αντιμετωπίσει την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε ούτε αρκετό χρήμα, αρκετούς πόρους. Το μόνο μέσο που υπήρχε ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκεί δεν έχουν πλειοψηφία τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν την πλειοψηφία. Και όλα τα κράτη-μέλη είναι μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από μόνο του, από μόνο του αν αναλάμβανε την υπόθεση, θα σήμαινε ότι θα εφήρμοζε παγκόσμιους κανόνες σε, κατα... σε αγορές. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ήταν σωστό να εφαρμόσουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Και έτσι καταλήξαμε στο μοντέλο της Τρόικα διαφορετικά θεσμικά όργανα, διαφορετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διαφορετική δημοκρατική νομιμότητα, αλλά ένα μέσο διακυβερνητικό και όχι κοινοτικό. Εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή θα ήταν αυταπάτη όπως ε, είπε ο Διευθυντής ε, του ε, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Στις ακροάσεις, στις αποστολές μας, το έχουμε δει αυτό. Σήμερα έχουμε προχωρήσει και έχουμε επιτυχία. Καμία χώρα δεν χρεοκόπησε, η Ευρωζώνη είναι σταθερή, δύο κράτη-μέλη, η Ιρλανδία και η Ισπανία μπόρεσαν ήδη να εγκαταλείψουν τα προγράμματα της, Τρόικα, της Τρόικας. Η ανάπτυξη ε, βελτιώνεται, έχει εφαρμοστεί η ρύθμιση για τις τράπεζες, έχει δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και ε, έχει μειωθεί η συμμετοχή της Τρόικας από το 1 τρίτο στο 10% των προγραμμάτων. Έχουμε λοιπόν τώρα περισσότερο χρόνο για την εφαρμογή των προγραμμάτων ε, και για την αποπληρωμή των χρεών. Ωστόσο, και κλείνω, πρέπει ως βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και ως Ευρωβουλευτές πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο διαφέρει η νομιμότητα, υπάρχει έλλειψη κοινών ελέγχων και λέγεται ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τις διαδικασίες και να εξάγει ε, συμπεράσματα, ενδεχομένως ε, να φτάσουμε και σε τροποποίηση ε, της συνθήκης. Και Θέλουμε επίσης διαρθρωτική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη και απασχόληση. Και γύρω από αυτά στρέφεται η έκθεσή μας και υποβάλλουμε προτάσεις για το μέλλον. Δεν απαιτούμε η Τρόικα να σταματήσει τις εργασίες της, πρέπει να ολοκληρώσει τα προγράμματα, αλλά θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Τρόικας. Και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εξάγει συμπεράσματα τα οποία να μπορέσουν να οδηγήσουν σε μελλοντικά μέτρα. Ελπίζω λοιπόν έτσι να έγινα σαφής και να κοιτάμε το μέλλον, αντί να προσπαθούμε να ρίξουμε ευθύνε για το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάρας. Να σας θυμίσω ότι Συμπροεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γιάννης Τραγάκης. Και συμπροεδρεύω κι εγώ ε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον άλλον συνεισηγητή της έκθεσης πρωτοβουλίας, τον ε, συνάδελφο Λιέμ Χουάν Γκότς, για 10 λεπτά. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη μόλις σας το είπε και ο Ότμαν άρρωστε. Είναι πολύ ευαίσθητη διότι σήμερα στην Ευρώπη αμφιβάλλουν όλοι για τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Τρόικας καταρχάς και κατά δεύτερον ο λαός σήμερα αμφιβάλλει κατά πόσον είναι αποτελεσματική η πολιτική που συστήνεται παντού. Όλοι μέχρι τώρα ήταν ερωτευμένοι με την Τίνα. Ε, ξέρετε ποια είναι η Τίνα. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση για αυτήν. Ακόμα και ο πρόεδρός μου, ε, ο πρόεδρος τη Γαλλία είναι ερωτευμένο μαζί τη. Αστειεύομαι φυσικά. Αλλά όπου και να δούμε την καθημερινή ζωή, κανένας δεν τη θέλει αυτή την Τίνα. Ακούμε λοιπόν όλη αυτή τη συζήτηση και ο κύριος Μπαρόζο επιμένει να εφαρμόζουμε την ίδια πολιτική, την ίδια μακροοικονομική πολιτική σε κάθε χώρα για να αντιμετωπίσουμε πόρο διαφορετικές καταστάσεις. Και αν συγκρίνουμε και τις τέσσερις χώρες ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουμε τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία. Η αγορά εργασίας εκεί είναι ευέλικτη δεν υπάρχει ανάγκη για διαρθρωτική αλλαγή στην αγορά εργασίας και η περίπτωση της Ιρλανδίας είναι η περίπτωση της τραπεζικής κατεξοχήν κρίσης. η οποία υποτίθεται ότι σήμερα θα επιληφθεί αναδρομικά μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας κάτι το οποίο δεν δέχεται κανένα μέλος κυβέρνησης. Εάν δεχτούμε την περίπτωση της Πορτογαλίας, εκεί δεν έχουμε τραπεζική κρίση, αντίθετα με την περίπτωση της Ιρλανδίας. Η περίπτωση της Πορτογαλίας έχει προκύψει από ε, ένα μεταδοτικό φαινόμενο της ελληνικής κυρίως κρίσης. Και αν δούμε την ίδια την Ελλάδα, Εάν το πρόγραμμα του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχε εφαρμοστεί νωρίτερα μαζί με άλλα μέτρα, μπορεί ίσως να μην είχαμε συνέπειες για την πορτογαλική οικονομία και για την κυπριακή οικονομία. Έγινε λοιπόν πολύ μεγάλη συζήτηση σε κάθε χώρα Και γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή και εντός της ίδιας της Τρόικα. Ακούμε τα μέλη της Τρόικα και από αυτά που μας είπαν διαπιστώσαμε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν απαραίτητο η ίδια με τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναφέρομαι στην όλη συζήτηση για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι δεν ήταν ε, ε, σωστός, ήταν ασθενής αυτός ο πολλαπλασιαστής και έπρεπε να είναι ισχυρή η θέση μας. Η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όμως όπως γνωρίζετε δεν ήταν η ίδια θέση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλεγε ότι οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές είναι υψηλοί και ίσως ε, υποτιμήσαμε και τις συνέπειες της ε, εξυγίασης, της δημοσιονομικής εξυγίασης. Η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν περισσότερο να γίνεται μια εσωτερική εξολόγηση και διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Και μετά Είχαμε και όλες αυτές τις συζητήσεις μεταξύ του λαού εντός των κρατών μελών, ε, είχαμε τις συζητήσεις μεταξύ των μελών της Τρόικας ε, και το θέμα είναι πού έγιναν όλες αυτές οι συζητήσεις ε, από εκεί και πέρα ε, και πού εξετάστηκε κατά πόσον το αντικείμενο των συζητήσεων αυτών ήταν ε, σωστό. Πουθενά. Και ποιες ήταν οι συνέπειες. Οι συνέπειες ήταν ότι η Τρόικα εφήρμοσε ίσως και υπερβολικά όλες τις περιοριστικές λύσεις ε, από μακροοικονομική σκοπιάς. Σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα από το πρόβλημα, γίνονταν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας. Σε κάθε χώρα υπάρχουν ισχυρά μέτρα εξυγίανσης του προπολογισμού. Κάθε χώρα έχει περιορισμούς και έχει περιορίσει τις ιδιωτικές και τις δημόσιες δαπάνες. Και οι συνέπειες τις ε, επισημαίνουμε και στην έκθεση είναι ότι οι στόχοι από μακροοικονομική σκοπιάς δεν έχουν επιτευχθεί. Βεβαίως βραχυπρόθεσμα η Τρόικα απέφυγε τη χρεοκοπία. Αλλά μακροπρόθεσμα, εάν δούμε τα στοιχεία για τις πιθανότητες ανάπτυξης, αν δούμε τα στοιχεία για την αναλογία ε, χρέους ε, ΑΕΠ και ιδίως αυτό το στοιχείο, η αναλογία χρέους ε, ΑΕΠ είναι πολύ υψηλότερο από ότι ε, πριν ε, εφαρμοστούν τα προγράμματα χρηματοοικονομικής βοήθειας. Και μετά, οι πηγές του προβλήματος δεν έχουν ξανεμιστεί, η κρίση δεν έχει τελειώσει και το θέμα είναι πώς μπορούμε να αποφασίσουμε για το ποιες είναι οι καλές λύσεις για το μέλλον. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να αποφασίσει είναι η δημοκρατία. Το γνωρίζετε γιατί είστε βουλευτές. Χρειάζομαστε τη δημοκρατία προκειμένου να αποφασίσουμε αν οι λύσεις αυτές ήταν καλές, και, ήταν ποιες θα είναι οι καλές λύσεις για το μέλλον. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στο τελευταίο τμήμα της έκθεσής μας, αναφερόμαστε στη δημοκρατία και, ο συνάδελφος και εγώ αναφερόμαστε στο μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Διότι αν δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ευρώπη, εμφανίζεται ο ευρωσκεπτικισμός. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένε προτάσεις. Και θεωρώ ότι η έκθεσή μας δεν έχει μόνο συμβαλικό χαρακτήρα, χρειάζονται και άλλες εκθέσεις, χρειάζονται και νομοθετικά μέτρα, χρειάζεται ίσως και αλλαγή της συνθήκης, όταν θα έχει οριμάσει βέβαια και ο χρόνος για να γίνει η αλλαγή. Τι εννοούμε πιο συγκεκριμένα. Θεωρούμε ότι ο μηχανισμός σταθερότητας είναι το πρώτο βήμα για την εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα υποκαταστήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση μέσω της κοινοτική μεθόδου. Αν θέλουμε να υπάρχει, θέλει να, ε, να υπάρχει δημοκρατική λογοδεσία. Το πρόβλημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τη σήμερα ημέρα είναι ότι είναι ένας ε, ε, διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά το βασικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσετε εσείς ως εθνικοί βουλευτές είναι αυτό το οποίο αποκαλεί η κυρία Μέρκελ μακροοικονομική αιρεσιμότητα και εμείς ε, την έχουμε βιώσει αυτήν. Μακροοικονομική αιρεσιμότητα χωρίς δημοκρατία σημαίνει προβλήματα. Μπορούμε σήμερα να έχουμε μακροοικονομική αιρεσιμότητα χωρίς να υπάρχει δημοκρατική λογοδοσία. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε αύριο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε με τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα. Και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, σιωπήσουν και δεν μπουν τίποτα για τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ε, θα αποφασιστούν με διακυβερνητικό τρόπο, θα βρεθούμε εμείς στις χώρες μας ενώπιον του ίδιου προβλήματος που αντιμετωπίζει η Τρόικα σήμερα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι συνταγές οι οποίες δεν κατάφεραν να λύσουν την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν και η έκθεση για την Τρόικα δεν είναι μία απλό συμβολική έκθεση, σηματοδοτεί το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε έτσι περαιτέρω, χρειαζόμαστε τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκότς. Και τώρα δίνω στο λόγο στον κύριο Λάμερτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, στο βαθμό που υπάρχει και όσο θα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητεί με αυξανόμενο αριθμό αυτή των κρατών, όχι μόνο για την διεύρυνση και εμβάθυνση της κοινή μας συνεργασίας, αλλά και για την δημοκρατική νομιμοποίησή της. Άρα στην Ευρώπη δεν μας ενδιαφέρει μόνο αν αυτό που κάνουμε όλοι μαζί είναι αποτελεσματικό, αν ε, χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αν βρίσκει αποδοχή, αλλά μας ενδιαφέρει επίσης πολύ αν όλα αυτά χαρακτηρίζονται από δημοκρατική νομιμότητα. Εκτός Ευρώπης αυτή η συζήτηση δεν γίνεται καθόλου ή γίνεται πολύ αργά και διστακτικά. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε περί ποιου θέματος ομιλούμε στα πλαίσια αυτής της προβληματικής. Θα έλεγα ότι με ενοχλεί λίγο το αυτονόητο ε, έλλειμμα, όπως το, το λέμε, στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει άλλος διεθνής οργανισμός που να τον βλέπω εγώ και να έχει τόση δημοκρατική νομιμοποίηση στις διαδικασίες που ακολουθεί ε, περισσότερο δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει το θέμα δημοκρατική νομιμοποίηση να μην είναι το μόνο που θα μας απασχολεί. Ε, αναφέρομαι και στο θέμα της έκθεσης των δύο συναδέλφων. Ας δούμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για προγράμματα βοήθειας, ε, για σειρά ε, κρατών μελών και δεν μιλάμε για ε, υποχρεώσεις με βάση την κειμένη νομοθεσία, αλλά για μέτρα που λαμβάνονται παρόλο που συμβατική υποχρέωση δεν υπάρχει. Και επειδή δεν υπάρχει βρέθηκε μια κατεξαίρεση λύση ειδική ώστε οι χώρες αυτές να βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Αυτό, ομολογουμένος, είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να επανεξετάζεται για να βλέπουμε εάν ε, επιτυγχάνονται οι στόχοι, αν ε, υπάρχει αποτελεσματικότητα, αν υπάρχει διαφάνεια, αν υπάρχει αποδοχή από τις χώρες και αν υπάρχει και δημοκρατική νομιμοποίηση πριν μιλήσω για την αποτελεσματικότητα, θα πω για την αποδοχή. Αυτά τα προγράμματα βοήθεια στα μνημόνια ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ισπανία δεν έγιναν αποδεκτά από την ευρεία πλειοψηφία. Για λόγους πληρότητας πρέπει να πω ότι η αποδοχή αυτή δεν υπάρχει ούτε στη Γερμανία για παράδειγμα. Δηλαδή μια νυφάλια ε, ματιά δείχνει ότι κανείς δεν είναι ικανοποιημένος. Η μεν θεωρούν ότι βρίσκονται από μια δυσάρεστη, κάτω από μια δυσάρεστη πίεση. Οι άλλοι θεωρούν ότι καλούνται να προσφέρουν περισσότερα από όσα θέλουν και οι δύο κατηγορίες κρατών παραπονούνται στους εκπροσώπους τους για την κατάσταση αυτή. Η συζήτηση πρέπει να γίνει. Είμαι υπέρ. Αλλά το, δεν δέχομαι ότι μέσα σε αυτά υπάρχει έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα προγράμματα, τα μνημόνια. Με συμφωνία όλων των συμμετεχόντων. Γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση. Και γι' αυτό όλοι συμφώνησαν ότι θέλουν να βρουν κοινή λύση, διότι αυτό είναι προς το κοινό συμφέρον. Δηλαδή να αποφευχθεί μια ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Ο κύριος Κάλαρας ε, το είπε αυτό όταν αναφέρθηκε στις κρίσεις δεκαετίας του 20 και 30. Θέλουμε κοινή λύση, γι' αυτό επειδή δεν υπάρχει υποχρέωση που να απορρέει από τις συνθήκες, χρειάζεται ειδική συμφωνία, την οποία και κάναμε. Με βάση αυτή τη συμφωνία θα έπρεπε να συμφωνηθούν προγράμματα βοήθειας για τις χώρες σε κρίση, τα οποία θα πραγματοποιηθούν αν συμφωνήσουν και οι ίδιες οι χώρες των προγραμμάτων με τις ιδιαίτερε αυτές συμφωνίες, αυτό έγινε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Πορτογαλικό και το Ιρλανδικό και το Ισπανικό, ε, έγιναν διαβουλεύσεις στα κοινοβούλια τους και συμφώνησαν. Στη Γερμανία, για τη χώρα μου μπορώ μόνο να μιλήσω, ε, η νομοθεσία τι προβλέπει. Επειδή η συμφωνία δεν μπορεί δεν μπορεί να λάβει συμφωνία χωρίς να ε, αποφανθεί και να συμφωνήσει και το Κοινοβούλιο. Ακόμα και αν υπάρχουν αλλαγές, τροπολογίες στη συμφωνία, πάλι θα πρέπει να συνδράμει το Κοινοβούλιο ούτως ώστε να έχουν νομική ισχύ. Έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας σίγουρα δεν υπάρχει λοιπόν. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι αν έχουν αποτελέσματα τα προγράμματα που προβλέπουν τα μνημόνια. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτυγχάνουμε αυτά που θέλουμε μέσα από τα προγράμματα, όπως τα είχαμε σκεφτεί. Εκεί είναι θεμητές οι αμφιβολίες, αλλά δεν είναι το θέμα η δημοκρατική νομιμοποίηση. Και τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις ακόμα ενίοτε σφάλουν ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το αποκλεί αυτό. Γι' αυτό ε, υπάρχει μια κοινοβουλευτική παρακολούθηση αυτών των διαδικασιών, ούτω ώστε οι υποθέσεις, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί να εξετάζονται και να αναθεωρούνται και να ε, αξιολογούνται με βάση τις εμπειρίες. Και θα μπορούμε να δούμε αν με βάση την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα από αυτό το ειδικό μόρφωμα, αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση που έχουμε, αν από αυτή μπορούμε να έχουμε μια, ένα μόνιμο μόρφωμα. Ε, εγώ Καταρχήν δεν θα σταθώ εμπόδιο σε μια τέτοια εξέλιξη. Θα ήθελα όμως να γνωρίζω αν εκτός από τις χώρες που έχουν το ευρώ ως νόμισμά τους και οι άλλες χώρες που δεν έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ, όχι ακόμα, οι άλλοι που δεν θέλουν ενδεχομένως ποτέ να το εισαγάγουν ως νόμισμα, αν όλες αυτές οι χώρες είναι διατεθειμένες να το εντάξουν αυτό το μόρφωμα στην ε, κειμένη νομοθεσία. Αν δεν διευκρινιστεί το θέμα αυτό, θα πρέπει να ζήσουμε με αυτά τα βοηθήματα, τα βοηθητικά μορφώματα και δεν θα πρέπει να γίνεται κριτική όλων ε, εναντίον όλων. Είναι αυτό το αποτέλεσμα της σημερινής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμπεριλαμβανομένων και των επιδιώξεων κάποιων κρατών σε ό,τι αφορά τη μελλοντική πολιτική τους. Τέλος, ε, θα ήθελα να αναφέρω κάτι ακόμα. Ελπίζω ότι κατέδειξα ότι το θέμα της ε, δημοκρατικής νομιμότητας, που θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να το συγχαίουμε με το θέμα της δημόσιας αποδοχής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας των μνημονίων. Και εγώ έχω την υποψία που, ότι τη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε για την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που είναι σύνθετα πρέπει να την διευκολύνουμε ε, επικεντρωνόμενη στο θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας που έχει λυθεί ενώ το θέμα της αποτελεσματικότητας των μνημονίων χρήζει μιας, μιας σε βάθος συζήτησης. Και αυτό με οδηγεί σε ένα άλλο θέμα σχετικά με τα τρέχοντα μνημόνια και την αποτελεσματικότητα και αποδοχή τους. Ε, εδώ πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις που έχουν, αλλά και τις παρεπόμενες ακούσιες επιπτώσεις και τις αντιρροπιστικές δράσεις που μπορεί να έχουν. Ε, επίσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν επανεξετάζονται μόνο οι προπολογισμοί των κρατών μελών, αλλά και υπάρχουν και ε, συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάθε χώρα ούτως ώστε να υπάρχει εξέλιξη στα κράτη-μέλη που θα ε, προωθεί το κοινό όφελος, ε, την εσωτερική αγορά και τις πολιτικές μας γενικότερα. Γίνονται συστάσεις λοιπόν για την οικονομική πολιτική των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα ότι και στα, Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προπάντων θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει, δεν το επικρίνω. Ε και προφανώς θα πρέπει να συζητούμε με βάση ετήσιες εκθέσεις πώς, εκτιμούμε την οικονομική συγκυρία, τις εξελίξεις, τα φορολογικά έσοδα, τι προβλέπετε, τι δαπάνες μπορούμε να κάνουμε χωρίς να ε, υπονομεύσουμε τις οικονομικές ισορροπίες, τι ε, βράχοι και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις θα υπάρχουν στους προϋπολογισμούς. Όλα αυτά που είναι αυτονόητα σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να γίνονται από κοινού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όχι μόνο δεν είναι επικριτέα μια τέτοια ε, προσπάθεια, αλλά είναι και ευπρόσδεκτη. Ε, με αυτές τις αιτήσιες ε, δημοσιονομικές, οικονομικές προοπτικές ε, και εκθέσεις έχουμε υψηλής προτεραιότητας σε πολιτικά προγράμματα. Αυτά που η Κομισιόν ή ο Επίτροπο υπεύθυνο για την εσωτερική αγορά ή ο Επίτροπο για τον προπολογισμό, αυτά που προτείνει η Κομισιόν και η Επίτροπη, είναι η υλοποίηση των προσδοκιών ε, για τι περαιτέρω εξελίξει, η εφαρμογή των προτεραιοτήτων και όλα αυτά είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένα, αλλά χρήζουν και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θεωρώ ότι αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, αυτά που συστήνει για τις χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν θεωρηθούν αυτά ως κοινή βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό εδώ βρίσκω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε ακόμα καλύτερα να διαχωρίσουμε τις εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του καθενός και να προχωρούμε σε κοινέ αποφάσεις. Βουλής και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ντόμινικ Χάνιγκαν, ε, πρόεδρο Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Uh, Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για την Ιρλανδία είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Πετύχαμε τους στόχους μας και καταλήψαμε το πρόγραμμα διάσωσης ε, τον προηγούμενο μήνα. Πριν δύο εβδομάδες ε, συγκεντρώσαμε τέσσερα δις ε, στην, στις αγορές με δημόσια χρεόγραφα. Σίγουρα λοιπόν αποτέλεσε επιτυχία το πρόγραμμά μας, έχουμε πάλι πρόσβαση στις αγορές. Την ε, προηγούμενη Παρασκευή η Moody's αναβάθμισε το, ε, ε, την, αξιο, την, την πιστοληπτική μας ικανότητα και η αδιαμφισβήτητη αυτή η οικονομική επιτυχία έχει αφήσει κάποιες κοινωνικές συνέπειες τις οποίες θα νιώθουν οι Ιρλανδοί για πολλά χρόνια στο μέλλον και είμαι βέβαιος ότι αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Θα ήθελα να αναφερθώ στο γιατί η Ιρλανδία έπρεπε να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Φορολογικές ελαφρύνσεις που εισήγαγε η προηγούμενη κυβέρνηση και περισσότερη ε, πρόσβαση σε πιστώσει ε, στις ε, ευρωπαϊκές τράπεζες οδήγησε σε φούσκα στα ακίνητα και έτσι αγορά πολλών κατοικιών. Μετά όμως κατέρευσε η Λέμαν Brothers και οι τράπεζές μας συνειδητοποίησαν ότι ήταν καταδικασμένες χωρίς εξωτερική βοήθεια. Έτσι λοιπόν ασκήθηκε πίεση στην κυβέρνηση όχι μόνο από τις τράπεζες αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και από άλλους που ανησύχησαν ε, σχετικά με τις συνέπειες για το ευρώ και άλλες οικονομίε. Και γι' αυτό οργανώθηκε γρήγορα ένα πρόγραμμα διάσωση. Η Ιρλανδία αναγνωρίζει απολύτω ε, την ε, εθνική μας ευθύνη στην κρίση αυτή, ωστόσο είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση και κοινή ευθύνη επίσης. Η Ευρώπη δεν είχε τότε τις πολιτικές επιλογές που έχει τώρα στη διάθεσή της, ε, δεν είχαμε την δυνατότητα του Μπέιλιν που έχει συμφωνηθεί τώρα και η προηγούμενη κυβέρνηση της Ιρλανδίας ε, θέλησε ε, οι κάτοχοι ομολόγων ε, να συμμετάσχουν στη διάσωση των τραπεζών, ε, αλλά αυτό εμποδίστηκε από την Τρόικα. Και σημαντικό να αποφευθούν οι συνέπειες για την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι λοιπόν διασώθηκε το... διασώθηκαν οι τράπεζες. Ε, η διάσωση αυτή όμως στήχησε σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ στους Ιρλανδούς φορολογουμένους. και ε, η σχέση ε, ΑΕΠ και δημοσίου χρέους είναι 120% σε σχέση με 80% που ήταν ε, πριν. Αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση μας άφησε ένα έλλειμμα 14% και με λογικά επιτόκια να χρηματοδοτήσουμε αυτά ήταν αδύνατον και γι' αυτό ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα μαζί με το, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι είχαμε πρόσβαση σε 85 δις ευρώ για να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας, θα μας ε, θα αποκαταστήσει την οικονομία μας και θα την κάνει βιώσιμη. Αυτό απέτησε φορολογικές αυξήσεις, ε, περικοπές, ε, πώληση κρατικής ιδιοκτησίας και μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Και προϋπολογισμοί λιτότητας κάθε χρόνο σημαίνουν ότι τώρα ε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο του ε, ε, ελλείμματος ύψου σε 3% και ισοσκελισμένου ε, ισοζυγίου και ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Έχουμε όμως αυξημένη φτώχεια, αυξημένη μετανάστευση και αυξημένο χρέος. Ε, ήταν ε, πολύ ε, χοντρό, αποτελεσματικό όμως το μέσο της Τρόικας. Πετύχαμε τους δημοσιονομικούς στόχους, δεν πετύχαμε όμως τους άλλους στόχους μας και το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Ναι, έγινε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, αλλά οι εθνικοί βουλευτές λίγα είχαν να πούν όσον αφορά το περιεχόμενο του μνημονίου. Ε, βρέθηκαν ε, πρώτε τελεσμένων. Και οι πολίτες ε, δεν είχαν καθόλου λέγει. Η πρώτη δυνατότητα που είχαν να εκφράσουν άποψη για οποιοδήποτε από τα ευρωπαϊκά μέτρα ήταν όταν εγκρίθηκε με δημοψήφισμα το σύμφωνο. Δεν, ένιωθαν όμως ότι δεν γίνονται αρκετά από την Ευρώπη στον μη δημοσιονομικό τομέα. Ε, και γι' αυτό χαιρόμαστε που επιτέλους υπήρξε συμφωνία για προβλήματα όπως είναι η εγγύηση για τους νέους, στο πακέτο απασχόλησης και επίσης επικροτούμε τις προτάσεις της Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση στην ε, ΟΝΕ. Κατά τη διάρκεια του, του προγράμματος ε, η Τρόικα δεν ε, εμφανίστηκε στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο παρότι είχαν ε, κατηδίαν συναντήσεις με βουλευτές. Ήταν προφανώς αποτυχία το ότι θα έπρεπε να συμμετάξει το, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε κάτι που ήταν εσωτερικό ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο συχνά καταλάβαινε καλύτερα τις συνέπειες της λιτότητας ε, και τι θα γίνει τώρα στο μέλλον. Όπως είπαμε, επιστρέψαμε στις αγορές, έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, η ανεργία μειώνεται κάπως. Αλλά εάν δεν δούμε ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει αναγνώριση της μοναδικής θέσης μας όσον αφορά ε, τα τραπεζικά χρέη, τότε ανησυχούμε αν θα είναι βιώσιμη η οικονομία μας και γι' αυτό θα ήθελα να επενέσω την, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής για την Τρόικα. Τώρα έχουμε χρόνο για μια ανάσα. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει οι διαδικασίες αυτές ε, να ε, ελέγχονται. Σίγουρα η δημοσιονομική πολιτική είναι ένας τομέας που απασχολεί πολύ τις ε, εθνικές κυβερνήσεις, αλλά ε, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει λέγει σε αυτά, εάν ελέγχει τις διαδικασίες μεταξύ Τρόικας, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τότε τίθεται το θέμα μήπως η περισσότερη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχει περισσότερα ωφέλη κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι προς συζήτηση, αλλά μπορούμε όλοι να συζητήσουμε ότι δεν είναι βέλτιστο το αποτέλεσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η Ιρλανδία και η Ελλάδα έχουν ε, ε, αναλογία χρέους προς ΑΕΠ άνω του 100% και ο Τζον Άνταμς είπε ότι υπάρχουν δύο τρόποι να κατακτήσει κανείς ε, ένα κράτος, ο ένας είναι με το σπαθί, ο άλλος είναι με τα χρέη. Κανένας δεν θέλει να δει μια Ευρώπη δύο ζωνών με ε, αφέντες και σκλάβους. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια. Η Ιλλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία μπορεί να είναι οι άτυχες χώρες σε αυτήν την ε, οικονομική κάμψη, αλλά μπορεί να είναι άλλες χώρες την επόμενη φορά. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να δείξουμε στον κόσμο ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι απλά μια ελπίδα, είναι κάτι που υπάρχει ήδη σήμερα. Ε, σίγουρα είχε καλές προθέσεις η βοήθεια που λάβαμε από την Ευρώπη, αλλά δεν ε, ανταποκρινόταν σε αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε λοιπόν ε, στήριξη προς τον ε, Ιρλανδό φορολογούμενο για να σταματήσουμε τις συνέπειες ε, για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και ε, γι' αυτό θέλαμε να ανακεφαλοποιήσουμε τις τραπεζές μας. Το μέλλον μας είναι κοινό και τώρα που οι οικονομίες μας βγαίνουν από την ύφεση θα πρέπει να εξετάσουμε τις ανάγκες της κάθε χώρας. Οι ιδρυτές της Ένωσης δεν ήθελαν μια Ευρώπη πλούσιων και φτωχών χωρών. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε τις ανάγκες μας ώστε αυτή η Ένωση Κρατών να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες. Να μην συνθλίβεται καμία χώρα από χρέη. Υπάρχουν εργαλεία στη διάθεσή μας όπως είναι το, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και η Τρόικα μας βοήθησε να κάνουμε τις επώδυνες προσαρμογές για να αποκαταστήσουμε την οικονομία μας. Αλλά μην πιστέψετε ούτε ένα λεπτό ότι επειδή μια χώρα εγκαταλείπει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ότι η χώρα αυτή είναι πάλι υγιής και σε καλή κατάσταση. Χρειαζόμαστε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να είναι βιώσιμο το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντόμινικ Χάνιγκαν, πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδικής Βουλής και δίνω το λόγο στον κύριο Αλεχάνδρο Θέρκας, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Τέσσερα λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο, κύριε Στέρκας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλώ εξ ονόματός μου, αλλά και εξ ονόματος των μελών ε, του Κοινοβουλίου της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, διότι θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι κάθε φορά που αναφερόμαστε στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Απασχόλησης αυτοπροσκλήθηκε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε και εμείς να κάνουμε μια έκθεση, εκπονούμε μια έκθεση για τις κοινωνικές συνέπειες ε, των ε, μνημονίων αυτών για τους πολίτες μας. Ε, ξέρουμε βέβαια ότι μπορεί να είμαστε λίγο ενοχλητικοί προσκεκλημένοι γιατί θα παρουσιάσουμε μια λίγο διαφορετική εικόνα από αυτήν που προσπαθούν να μας πλασάρουν αυτές τις μέρες ότι αυτά τα μνημόνια ήταν σαφή, ξεκάθαρα και ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση. Και ε, μάλιστα, όπως είπε και κάποιος από τους προλαλήσαντες, έγιναν ε, και δημιούργησαν ένα καλύτερο κόσμο. Δεν είναι αυτή η καθημερινότητα των πολιτών. Διαβουλευθήκαμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, μιλάμε τα πανεπιστήμια, υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση στο Κοινοβούλιο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τεκμηρίωση που μας παρουσιάζει μια πραγματική κοινωνική καταστροφή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κλαμπ τραπεζιτών, ούτε ένα κλαμπ ε, τεχνοκρατών, αλλά είναι μια δημοκρατική δομή για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς και δεν θα πρέπει να λησμονούμε τους πολίτες μας. Το άρθρο 9 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι όλες οι πολιτικές και όλες οι δράσεις στόχο έχουν να επιτύχουμε υψηλό ποσοστό απασχόλησης και υψηλό ποσοστό κοινωνικής ένταξης. Και κυρίες και κύριοι, ε, αυτά με βάση τη συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση στι τέσσερι χώρε είναι είναι μια κοινωνική καταστροφή. Καταστράφηκαν όλες οι κοινωνικές δομές. Σε λιγότερο από τρία χρόνια έχει ε, φτάσει στα ύψη ανεργία και μάλιστα έχει σταματήσει και η παραγωγή. Σε μια χώρα μειώθηκε και 25% η παραγωγή. Υπάρχει μαζική μετανάστευση νέων στην Ιρλανδία και στην Ισπανία. Χάνεται μια ολόκληρη γενιά. Έκλεισαν νοσοκομεία. Χάσουμε του στόχου Ευρώπη 2020 και πραγματικά έχουμε οπισθοδρομήσει σε όλου του μεγάλου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κύριε και κύριοι θα πρέπει κάπου να τα γιατί αυτή είναι η καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών των χωρών του Νότου που έχουν χάσει τι θέσει εργασία του, έχουν χάσει τα δικαιώματά του. Το 70% των Πορτογάλων εργαζομένων που είχαν συλλογικές συμβάσει πλέον δεν εργάζονται με βάση συλλογική σύμβαση. Και ξέρω ότι αυτή είναι μια εικόνα που δεν σας αρέσει, διότι εσείς δεν έχετε καμία κοινωνική ευαισθησία. Αλλά οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν κοινωνική ευαισθησία. Και όταν κάποιος αναρωτιέται γιατί οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή απορρίπτουν αυτή την πολιτική της Τρόικας, ε, ίσως η Κεντρική Ευρώπη δεν το αντιλαμβάνεται, διότι δεν έχετε δει τι συμβαίνει στους δρόμους, τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις. Ρωτήστε τους εκατοντάδες χιλιάδες ε, Ισπανούς επιχειρηματίες που έχουν ε, κλείσει γιατί δεν έχουν ε, πιστώσει δεν έχουν δανειοδότηση και πρέπει να πληρώσουν πολύ υψηλότερα επιτόκια από του Γερμανού επιχειρηματίε. Ή ρωτήστε ένα νέο Ισπανό που έχει πέντε φορέ λιγότερε πιθανότητε να βρει μια θέση εργασία από ότι ένα άλλο Βορειοευρωπαίος. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιος μια κοινωνική καταστροφή που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική καταστροφή και πρέπει εμεί να αναστρέψουμε την κατάσταση. Ε, τέσσερα λεπτά έχω χρόνο να μιλήσω αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, πρέπει να κάνουμε μια πραγματική μελέτη όλων των συνεπειών, όπω έλεγε χθε ο κύριο Μπαρόσο και όπω έλεγε ο κύριο ε, Ότμαν Κάρα σήμερα Όλε τι συνέπειε. και το τι συμβαίνει στην καθημερινή ζωή, όχι μόνο την υγεία των τραπεζών, την υγεία των οικογενειών, των πραγματικών επιχειρήσεων και τη πραγματική οικονομία. Πρέπει να μελετήσουμε ει βάθος τι συνέβη για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη και στο μέλλον. Και θα πρέπει να ανακτήσουμε αυτά τα οποία χάθηκαν, διότι υπήρξε ένας διαρθρωτικός κίνδυνος, ο οποίος κατέστρεψε την οικονομία, την παιδεία, τη φτώχεια. Και πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη ε, και να δούμε, διότι αν δεν υπάρχει απασχόληση, αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να διασώσει το νόμισμά της. Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να διασώσει την οικονομία της, δεν θα διασώσει την κοινωνία της και θα χάσει το όραμά της. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Στέρκας ήταν εισηγητής της έκθεσης απασχόλησης και για τις κοινωνικές επιπτώσεις και του ρόλου της λειτουργίας της Τρόικα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. 13 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ αυτών. Επομένω, μπορείτε να λάβετε το λόγο. Κύριε Λάγκερ, πρέπει να συμπληρώσετε την κάρτα σας και θα σας δώσουμε το λόγο. Να ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση, να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε 4 ή 5 εθνικούς βουλευτές, έναν ευρωβουλευτή και χρόνο ομιλίας δύο λεπτά για τον καθένα με την συνάδελφο σκεύη κουκουμά ε, από την κύπρο. έχει το λόγο για δύο λεπτά. κυρία πρόεδρε ε, θα ήθελα να αναφερθώ στις διαδικασίες αποφάσεων και τη δημοκρατική νομιμοποίηση της τρόικας και να παραδεχτούμε όλοι ότι δεν πρέπει να δείχνουμε έκπληκτοι. η απουσία διαβουλεύσεων με τα συνδικάτα και τα κοινοβούλια η απουσία κάθε δημοκρατικού ελέγχου και κοινωνική λογοδοσία δεν είναι ανεξάρτητη από το διαχρονικό και εγγενέ δημοκρατικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση. και αυτό το έλλειμμα δεν είναι αφηρημένο. δεν υπάρχει άλλο τρόπο να περάσουν τέτοιε αντιλαϊκέ και βάρβαρε πολιτικέ παρά με τη φήμωση των λαών την καταστολή λαϊκών αγώνων όπου αναπτύσσονται και βέβαια με την παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην τοποθέτηση ενός από τους εισηγητές ότι δεν υπάρχει έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας στα προγράμματα που εφαρμόζονται. Να θυμίσω ότι και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η εισβολή και η κατοχή γινόταν με στρατιωτικά μέσα. Τώρα γίνεται με οικονομικά μέσα. Συμμεριζόμαστε το αίτημα να βρεθούν τρόποι για να καταστεί υπόλογη η Τρόικα και να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία των προγραμμάτων διάσωσης. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία, έστω και καθυστερημένα, από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής να επισκεφτεί τις χώρες και να αξιολογήσει τον ρόλο και τη λειτουργία της Τρόικας και αναμένουμε ότι θα καταγράψουν τις δραματικές συνέπειες σε όλες τις διαστάσεις και τις οικονομικές και τις ε, κοινωνικές που είχαν οι πολιτικές τους παρακολουθούμε μάλιστα τη συζήτηση που ξεκίνησε για πιθανή υποκατάσταση τη τρόικα από έναν ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. δεν είναι αυτό το ζήτημα το άμεσο αίτημα των λαών της Ευρώπης είναι να καταργηθούν οι πολιτικές αυτές και να ανατραπεί το περιεχόμενο και οι δυσβάσταχτες συνέπειες τους και όχι να αλλάξει το όχημα με το οποίο προωθούνται και επιβάλλονται. Ούτε πρέπει να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση στο πώς θα νομιμοποιηθεί θεσμικά η βαρβαρότητα των μνημονίων και η συνολική κοινωνικο-οικονομική πορεία της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Κουκουμά και ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο ε, Κάσο από το Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλή των Κοινοτήτων, για δύο λεπτά. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια πληττόμεθα και εμείς από τις δράσεις της Τρόικα και τις υπαγορεύσεις της και τα bailout και τις τραπεζικές προτάσεις, τις διασώσεις. Και βεβαίως ε, είναι σημαντικό να δούμε αν είναι δημοκρατικές και αποτελεσματικές. Πολλές φορές ε, είχαμε αντιδράσεις αλλά και ανεργία που αποσταθεροποίησε την Ένωση συνολικά. Όταν ο κύριοι Κάρας και Μπαρόσο αναφέρονται σε κοινωνικές επιπτώσεις, εγώ θα ήθελα να γνωρίζει ο κόσμος και να θυμάται ότι τα κοινωνικά θέματα έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και τον αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα στους εκλογείς αν δεν είναι ε, δημοκρατικά και αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δώσει στα εθνικά κοινοβούλια και στους εθνικούς εκλογείς, στο εκλογικό σώμα, μεγαλύτερο λόγο για να μπορούν να ανατρέπουν τις θέσεις σας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που όλο και περισσότερο θεωρεί ότι είναι το μοναδικό κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε νομίζω ότι θα συνεχίσει να επιδεινώνεται η κατάσταση και θα ανέλθει η άκρα δεξιά και επίσης θα έχουμε και πολύ αρνητικές συνέπειες ε, κατά τις ε, ευρωεκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάσου. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Ντανιέλ Λερουά από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι δύο συνάδελφοι, με τα οποία συμφωνώ για το ρόλο της Τρόικας, για τα συνέπειες για τις κοινωνικές συνθήκες. Ο συνάδελφος εξήγησε πολύ καλά ότι αυξήθηκε η φτώχεια στην Ιρλανδία και θεωρώ ότι το πρώτο στοιχείο θα ήταν να διευκρινίσουμε αυτή τη συζήτηση για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και ε, να δούμε τι γίνεται στα μνημόνια τα οποία συμφωνήθηκαν με τις χώρες για την οικονομική αναδιάρθρωση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, μια δογματική θεώρηση των πραγμάτων όπως έκανε η Τρόικα υπάρχει ε, οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος αναγνώρισε ότι υποτιμήθηκαν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές, ότι έκανε λάθος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ότι από το 2010 και τούδε ε, προσάρμοσε τους πολλαπλασιαστές σε κάποια προγράμματα. Η Τρόικα όμως δεν άλλαξε τα πράγματα, ε, συνέχισε σαν να μην είχε γίνει λάθος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε διαφάνεια και να ζητήσουμε να υπάρχει λογοδοσία για τα θέματα αυτά. Αν θέλουμε να έχουμε υποστήριξη στην ε, ανάπτυξη, δεν πρέπει όλα αυτά να είναι υποχρεωτικά οπωσδήποτε και θα πρέπει να πάμε λίγο πιο ήπια. Θα πρέπει το Eurogroup να είναι πιο επαγγελματικό και αυτά τα οποία μας είπε ο εισηγητής ε, δεν μας καθησυχάζουν σε καμία περίπτωση. Η δημοκρατική νομιμοποίηση θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα και θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση των κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η Τρόικα θα πρέπει να λογοδοτεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε όπως έλεγε ο Μολιέρος, ε, να ε, μην είναι ε, η κατάσταση, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Εντουάρτο Γκαμπρίτα από την Βουλή της Πορτογαλίας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Πορτογαλία είχε στον 20ο αιώνα την μακρότερη δικτατορία στην Ευρώπη και γι' αυτό η αλληλεγγύη, η δημοκρατία και η ανάπτυξη είναι για μας τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης. Στην Πορτογαλία μέχρι τώρα ε, δεν υπήρχε κόμμα που ήταν κατά της Ευρωπαϊκής ε, Ενοποίησης υπήρξαν αριστερές, δεξιές δυνάμεις, όχι όμως ευρωσκεπτικιστές που τάσσονταν κατά της, Ευρω... Ευρώπης. Το 2007 ε, και τώρα είχε 62% ε, ε, ε, χρέος και 3% έλλειμμα και μετά ε, πέρασε στην κρίση. Το μοντέλο της Τρόικας είναι ότι ασκήθηκαν, σημαίνει ότι ασκήθηκαν πιέσεις ε, στην ε, Πορτογαλία που οδήγησαν σε αμφιβολίες για, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καθυστερημένη απόκριση, αντίδραση της Ευρώπης ο καθυστερημένος χειρισμός θεμάτων ε, που ε, ήταν σαν να αντιμετωπίζαμε ε, ηθικά προβλήματα, δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες του λαού. Ακόμα και χθες όταν συνοψίστηκαν τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, αυτά περιορίστηκαν σε επιπτώσεις στην αγορά. Ε, δεν λήφθησαν υπόψη οι αναπτυξιακές ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι υπήρξαν θετικά αποτελέσματα στην Πορτογαλία σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, αλλά οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι σοβαρότατες. Οι επικείμενες ευρωεκλογές αποτελούν πρόκληση για την Ευρώπη που πρέπει να αποδείξει ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι εγχείρημα αλληλεγγύης, δημοκρατίας, νομιμότητας και ανάπτυξης. Η εναλλακτική είναι να συνεχίσουμε αυτήν την κίνηση προς τα ακραία αντιευρωπαϊκά κινήματα, ενώ η οικονομία καταραίει. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Τούσας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά για ένα λεπτό έχουν το λόγο οι ομιλητές για να απαντήσουν και να σχολιάσουν τις παρεμβάσεις. Κύριε Τούσα. Η διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια στα πλαίσια του Δημοσιονομικού Συμφώνου για την πορεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης όχι μονάχα δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά προβλήματα, τις αγωνίες και τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά και τις αντιστρατεύεται ανοιχτά. Τόσο κατά τη χθεσινή ημέρα από τους εκπροσώπους των ευρωνοσιακών οργάνων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κατά την σημερινή ημέρα από τους κεντρικούς εισηγητές επιβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα της συνέχισης με μεγαλύτερη ένταση της αντιλαϊκής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020 με στόχο την παραπέρα μείωση της τιμής εργατικής δύναμης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Πραγματικός στόχος και αυτής της διακυβερνητικής διάσκεψης είναι να δώσουν ψευτοδημοκρατική νομιμοποίηση σε όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Στη χειραγώγηση των λαϊκών συνειδήσεων για τον εξοραϊσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της καθώς και της αντιλαϊκής πολιτικής της που προωθείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα αν είναι σε διαδικασία μακροοικονομικής επιτήρησης ή μνημονίων. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην τραγική κατάσταση που είναι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας, αλλά θα αναφερθώ στην ατμομηχανή, την οικονομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 12 Σύμφωνα με τα επίσημα γερμανικά στοιχεία, 12 εκατομμύρια Γερμανοί ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ανεργία είναι της τάξης των 2.930.000. Το εισόδημα, το κατώτερο εισόδημα των Γερμανών εργαζομένων είναι 956 περίπου ευρώ. Άρα καλούμε μια, για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν την ίδια τους την πείρα να κλιμακώσουν τους αγώνες τους για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής Ευχαριστώ πολιτικής. Να ανοίξει ο δρόμος για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στην εξουσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τούσα. Uh, Κάποια πρώτα σχόλια από το μέλη του πάνελ. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Λάμπερτ. Ich möchte noch einmal... Θα ήθελα να πω ότι πρέπει όλοι να ενθαρρυνθούν να συζητήσουν για πράγματα που αξίζουν τον κόπο και έχουν νόημα. Όχι για θέματα που ουσιαστικά δεν αλλάζουν τίποτα. Βεβαίως και χρειάζεται αντιπαράθεση μεταξύ μας σχετικά με το αν τα μνημόνια εκπληρούν τους στόχους τους, εάν ε, συνδέονται με επιπτώσεις και παρεπόμενες επιπτώσεις που θέλουμε που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας ή όχι. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι τα τωρινά μνημόνια είναι τα μόνα δυνατά. Θα μπορούσαν να υπάρξουν κι άλλα, εναλλακτικά. Εμείς μιλάμε για αυτά που έχουν, είχαν συμφωνηθεί. Και ο σκοπός μιας τέτοιας συζήτησης ακριβώς αυτό συνίσταται σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πραγματική επίπτωση των προγραμμάτων. Δηλαδή, δημοσιονομικά, οικονομικά έχουν ε, την επίδραση που θέλαμε ή έχουν προβληματικές παρεπόμενες επιπτώσεις ε, που μας φαίνονται απαράδεκτες παρόλο που μπορεί να σταθεροποιούν τον προϋπολογισμό. Η αντιπαράθεση έχει νόημα πάνω σε αυτά τα θέματα. Και προφανώς αυτό είναι το καθήκον και των Εθνικών Κοινοβουλίων και των, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ποιο θα μας εμποδίσει να κάνουμε την αντιπαράθεση αυτή. Αλλά να μην ε, ε, κάνουμε σαν να μας ε, εμποδίζουν σκοτεινές δυνάμεις να ασκήσουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμερ και τώρα ο κύριος Χάνιγκαν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς θα αυξηθεί η λογοδοσία της Τρόικας. Εκφύσεως τα μέτρα ε, θα είναι δύσκολα και οδυνηρά σε οποιαδήποτε χώρα. Οι εθνικοί ε, βουλευτές θα επιχειρήσουν βέβαια να κατηγορήσουν την Τρόικα λέγοντας ότι εκείνοι τα λένε όχι εμείς, εμείς πρέπει να υπακούσουμε. Είναι δύσκολο να γίνει μια ε, σοβαρή και αποτελεσματική συζήτηση μεταξύ Τρόικας και ε, βουλευτών κατά τη ε, διάρκεια των μνημονίων. Γιατί θα κατηγορείται πολύ η Τρόικα. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να ε, αποδείξουμε ότι λογοδοτούν γιατί παίζουν ε, ρόλο και υπησέρχονται εδώ πολλά συμφέροντα ε, και σε επίπεδο ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ πολύ. Οι συνεισηγητές τώρα. Αυτή τη φορά πρώτα θα λάβει το λόγο ο Λίεμ Γκότς. Συνάδελφοι, τι θα ήταν διαφορετικό εάν τα κοινοτικά μέτρα θα είχαν εφαρμοστεί με λογοδοσία της Τρόικα. Ένα παράδειγμα να δώσω για να απαντήσω στον συνάδελφο Χάνιγκαν. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας υπήρχε ένα πρόβλημα με την Κεντρική τράπεζα. Το ξέρουμε αυτό, έχει γίνει σχετική συζήτηση. Ή μάλλον δεν έγινε συζήτηση ανάμεσα στην ε, Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχετικά με την ε, λύση που προτάθηκε. Το bail-in ή το bail-out, η εξωτερική διάσωση ή η εσωτερική εάν είχαμε την κοινοτική μέθοδο, ίσως να είχε επιλεγεί το Μπέιλιν, Η εσωτερική διάσωση, να φέρουν δηλαδή και οι ίδιοι οι μέτοχοι ε, το βάρος. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, κάνει άλλα πράγματα από το να ασκεί ε, η δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο αυτό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πολύ σοβαρό ερώτημα και στην περίπτωση της Ελλάδας μπορούμε πάλι να θέσουμε πιτάπιτο στο θέμα. Ε, έχουμε το λεγόμενο φαινόμενο τράγκη ε, και αυτό δεν έχει συζητηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λία Μότμαρ. Είναι πολύ λεπτό το θέμα και όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλον διότι υπάρχουν ε, διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές αρμοδιότητες, διαφορετικές αιτίες και διαφορετικά αποτελέσματα. Πολλά από τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε εκφράσεις οργής. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και τι μορφή έχουν αυτές. Όταν μια χώρα δεν μπορεί να προσφύγει στις αγορές ε, για χρηματοδότηση, για να χρηματοδοτήσει τα κοινωνικά, την εκπαίδευση, την υγεία, όταν δεν μπορεί να βρει χρήματα για ανάπτυξη και επενδύσεις, τότε χρειάζεται ένας μηχανισμός ώστε να μπορούν να ασκηθούν αυτές οι λειτουργίες. Και χρειάζεται χρόνος για να γίνουν ε, οι σχετικές προσαρμογές ε, και μεταρρυθμίσεις. Αυτό αναφέρθηκε από τον κύριο Λάμερτ. Πρόκειται για μια λύση ανάγκης, ε, μια προσωρινή λύση. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, χρειαζόμαστε μια μόνιμη λύση και τι μορφή θα έχει αυτή. Μια μόνιμη λύση είναι δυνατόν να υπάρξει με βάση το κοινοτικό δίκαιο ή θα πρέπει να είναι διακυβερνητική. Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά όργανα, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Αυτές είναι οι προσπάθειες που καταβάλουμε. Καταβάλουμε προσπάθειες για να διεξαχθεί ακριβώς αυτή η πολιτική συζήτηση και στην ε, Κοινωνική Επιτροπή και η ε, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ε, εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Θα πρέπει να συζητήσουμε τα ουσιαστικά ζητήματα για να δώσουμε μια σωστή απάντηση για το μέλλον να έχουμε λιγότερες παρεξηγήσεις και όταν μιλάμε για δημοκρατική νομιμοποίηση θα πρέπει να δούμε τα μέτρα πώς προετοιμάστηκαν, πώς εφαρμόστηκαν, πώς συμμετείχαν τα κοινοβούλια. Το θέμα δεν είναι απλά θεσμικό, έχει να κάνει με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος μετράει. Ε, τον κύριο Κάρας και τώρα το λόγο έχει ο Λόρδος Χάρισον, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Λόρδων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Uh, President, can I remind... Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επενθυμίσω στο συνάδελφο, στον Πιλκάς, ότι οι διαδηλώσεις στους δρόμους ήταν στο Κίεβο, διότι η Ουκρανία ήθελε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι να φύγει. Η Κροατία εντάχθηκε πέρσι και η Λετωνία εντάχθηκε προσφάτως στο ευρώ γίνεται μια έρευνα στη Βουλή των Λόρδων για τη βελτίωση της δημοκρατικής συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όχι για να είναι αντίπαλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά για να μοιράζονται από κοινού αυτά τα καθήκοντα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφο Ντόμινικ Χάνιγκαν να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θεωρείτε ότι πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτά τα οποία κάνουν τα, Ευρω... τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, για τη λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε ότι αυτό θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό σε σχέση με τις σχέσεις μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τις σχέσεις μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αφού αναφέρθηκε η Τρόικα σήμερα το πρωί, θεωρεί ότι η Τρόικα έχει εσωτερικές μεθόδους ε, σχέσεις και συνεργασίας μεταξύ των μελών της, διότι ε, κάποιες στιγμές φάνηκε ότι ερίζουν οι απόψεις εντό της Τρόικας. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συνεισηγητές τώρα, τον κύριο Κάρας και τον κύριο Χουαν Κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη βουλή εθνικών βουλευτών. Τι άποψη έχουμε γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η πρόταση και το θέμα είναι ε, πώς θα μπορεί να προέχει ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει τη φυσική του θέση ε, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, έχω να ρωτήσω το εξής. Μετά από τις επόμενες ευρωεκλογέ, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπάρχει ε, μια ξεχωριστή επιτροπή για την Ευρωζώνη. Εμείς που δεν συμμετέχουμε στην Ευρωζώνη, ε, θα ανησυχούσαμε ιδιαίτερα αν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι ως τα 28 μέλη της ενίας αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Λόρδο Χάρισον. Το λόγο έχει ο, Μπρούνο, ο κύριος Μπρούνος Μορόσμαν της Επιτροπής Προπολογισμού από το Αυστροϊακό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αφαιρθώ στον κύριο Λάμερτε και να πω ότι διαφωνώ στα όσα είπε για την νομιμοποίηση. Γιατί η είναι ένας θεσμός που δημοκρατικά δεν έχει νομιμοποιήσει και αυτό επηρεάζει την στρατηγική καταπολέμηση της κρίσης που πήγε να εφαρμόσει η Τρόικα στις αντίστοιχε χώρες και δεύτερον επηρεάζει και την πίεση που έπρεπε να ασκηθεί ώστε η ε, στρατηγική αυτή η νεοφιλελεύθερη να εφαρμοστεί στις χώρες. Σωστό είναι ότι ε, ψήφισαν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σωστό όμως είναι επίσης ότι υπήρξαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες ακριβώς ενάντια στα μέτρα αυτά και ενάντια στη συγκεκριμένη στρατηγική κατά της κρίσης διότι ε, συρρυκνώθηκαν ε, κοινωνικά προγράμματα, η πίεση ήταν μονόπλευρη διότι ε, υπονομεύθηκαν οι διαδικασίες ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυτό οδήγησε σε αντίδραση και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Επίσης, ε, σε αυτές τις χώρες δεν υπήρξε στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης. Βλέπουμε να αυξάνεται στις χώρες αυτές η ανεργία, εξακολουθεί να αυξάνεται η ε, ανεργία, άρα η κοινωνική συνοχή ε, θα πληγεί. Επίσης, ε, τα μνημόνια ασχολήθηκαν κυρίως με τη διάσωση των τραπεζών και όχι τη διάσωση του λαού, που αφέθηκαν στην τύχη τους. Και, κύριε Κάρας, αν θέλετε να κάνετε συγκρίσεις με τη δεκαετία του 30, αλήθεια είναι ότι ορισμένα έγιναν σωστά, αλλά δεν ε, λάβαμε υπόψη μας το New Deal του Roosevelt, δεν λάβαμε υπόψη μας την αυξανόμενη ανισότητα στην κατανομή εισοδημάτων και πλούτου. κυρία Μπάρμπαρα Λέτσι, της Επιτροπής Προεπιλογισμού της Ιταλικής Γερουσίας. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι πρέπει να αξιολογήσουμε αν νομιμοποιείται ή όχι, αν πρέπει να αυξήσουμε το δημοκρατικό έλεγχο στις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρώπη και οι οποίες εκχωρούνται στη συνέχεια στην Τρόικα, διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση. Όπως έλεγε και ο συνάδελφος από την Ευστρία προηγουμένως, ίσως θα έπρεπε να ενημερώνονται πάντα και καλύτερα όλοι οι λαοί οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε μια κατάσταση απόλυτης ένδυας. Ε, Υπάρχει βοήθεια η οποία ε, στοιχίζει όλο και περισσότερο στους απλούς ανθρώπους ε, προς όφελος των τραπεζών. Προσπαθούμε εδώ και τόσα χρόνια να τις ανακεφαλαιοποιήσουμε και φαίνεται ότι οι τράπεζες δεν κάνουν καν στη δουλειά τους στην Ιταλία ε, πλέον ο, ο λαός και η χώρα έχει λυγίσει εξαιτία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Και φαίνεται ότι δεν ε, είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να ελέγξει ούτε καν τι κάνει η κυβέρνησή μας. Εδώ και κάποιες μέρες έχει περάσει αυτό το νόμο για τη σταθερότητα, ένας νόμος ο οποίος εγκρίθηκε και ε, στηρίχθηκε σε δείκτες οι οποίοι είναι απόλυτα λανθασμένοι. Μας δείχνει μια ανάπτυξη άνω του 1%. Δεν υπήρχε έγκριση από κανένα Ινστιτούτο για αυτή τη μελέτη. Και όλα αυτά για να υπάρχουν περισσότερα έσοδα εις βάρος των πολιτών, να υπάρχουν ε, τραπεζικές εξηγιάνσεις και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν έλεγχο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και το τούπακ, η βιβέσμη των δύο μέτρων, ε, και φαίνεται ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τυφλή, διότι δεν ζητά ούτε τα απλά από την Ιταλική κυβέρνηση να κάνει μία αναθεώρηση των ιστορικών δαπανών. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Ιταλική κυβέρνηση, αντί να συνεχίσει να επιβάλλει στους πολίτες ε, να επαναλαμβάνει τα ίδια ασφάλεια, ασφάλματα, είτε είναι της Τρόικας, είτε είναι της Ευρώπη, είτε είναι της ε, Ιταλική κυβέρνηση εδώ και 20 χρόνια. Η το λόγο έχει τη Ροζάνα Αρτουρία από τη Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η απουσία ανάπτυξη και η μαζική ανεργία που βιώνουμε διακυβεύει την ε, μακροοικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η κρίση χρέους ε, διακυβεύει επίσης και την πολιτική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Εδώ και 10 χρόνια το ευρώ ουσιαστικά προκάλεσε γενική αναισθησία. Αναισθησία των αγορών, αναισθησία των ε, οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων. Και όταν ξέσπασε η κρίση χρέους, συνειδητοποίησαμε ότι πρόκειται για συστημική κρίση και χρειάστηκε να ε, σκεφτούμε κατεπηγόντως κατάλληλες λύσεις και ουσιαστικά να συσταθεί η Τρόικα. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η Ευρωζώνη δημιουργούσε μια πολύ συγκεκριμένη οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης. Όταν χρειάστηκε να δημιουργηθεί ένας ε, ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητος, οι εθνικές ε, ε, οικονομίες είναι αυτές οι οποίες χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν και όχι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια χρηστή διακυβέρνηση, οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση, οι οποίες θα συσταθούν βαθμιδών. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός σταθερότητας αλλά θα πρέπει να υπάρχει ε, και μια, ε, ένας υπουργό Οικονομικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ καλό να υπάρχει μία μόνιμη εποπτεία ε, έσω μίας επιτροπής η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των κοινοβουλίων των εθνικών κοινοβουλίων της Ευρωζώνης αλλά και ευρωβουλευτών. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια δημοκρατική νομιμοποίηση στην όλη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ε, διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και φυσικά αυτό θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη όσα μας προσφέρει το άρθρο 13 της ε, συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση. Θεωρούμε ότι η διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη θα πρέπει ε, να καταλήξει σε ένα ψήφισμα, αυτό σας προτείνω κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρτουρή και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λάγκεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο μετά τον κύριο Σάρκας, από, ε, τον Ευρωβουλευτή από την Ισπανία, που αναφέρθηκε στι στις ισπανικές εξελίξεις, που δεν είναι αντικείμενο της έρευνας της έκθεσης, ένα αυτό. Δεύτερον, τώρα, λίγο πριν από τις ευρωεκλογέ θα περίμενα πιο πολύ αυτοκριτική από τους συναδέλφους. Θυμάμαι πολύ καλά την οκταετία Σαπατέρο, και την Ισπανική Προεδρία, όπου ο κ. Σαπατέρο στην, ε, στο Ευρωκοινοβούλιο μίλησε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον ε, γάμο μεταξύ ομοφύλων. Αυτές ήταν οι, πρωτο, οι προτεραιότητές του. Ενώ ε, είχε αρχίσει για τα καλά η κρίση. Στη Γερμανία, με ο μεγάλος συνασπισμός έθεσε κάποιες προτεραιότητες αναγνωρίζοντας και ξεπερνώντας ε, ε, την κρίση. Λείπει η αυτοκριτική εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς. Η τραπεζική χρηματοπιστωτική κρίση ήταν το σημείο κινήσεως της κρίσης, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι σε όλες τις χώρες που υπήρχαν προβλήματα μέχρι την ε, χρηματοπιστωτική κρίση ήταν σοσιαλιστικές ε, σοσιαλιστικά κόμματα στις, ε, στην κυβέρνηση και στην Ισπανία και την ε, Πορτογαλία και την Ελλάδα και την Κύπρο και την Ιρλανδία, τη χώρα αυτή τη συγκρουσιακή. Και στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Ξέρω. Ξέρω, ξέρω. Ήταν κομμουνιστής ο πρόεδρος στην Κύπρο. Ναι, αλλά εδώ δίνεται μια μάχη για να τα λέμε σωστά. Δεν μπορούμε να παίρνουμε με απόλυτους όρους ένα μοντέλο. Και αν η Τρόικα ε, επιφορτίζεται από την Ευρωζώνη, τότε αναλαμβάνει μια εντολή. Εκεί που κάνω εγώ κριτική είναι στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν φρόντισε από πριν να αρθούν τα κακό κείμενα, να τηρηθεί το κοινοτικό κεκτημένο, να ελέγχεται η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, των διαρθρωτικών κονδυλίων. Στην περίπτωση της Ελλάδας που ήταν ιδιαίτερη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, διέθεσε έναν επίτροπο που θα αναλάμβανε και θα ήταν υπεύθυνος για την Ελλάδα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν διατεθειμένη ε, κάποιους ε, ε, Έλληνες συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τους στείλουν για να βοηθήσουν να βελτιωθεί και να μεταρρυθμιστεί η δημόσια διοίκηση, διότι υπάρχουν υψηλής εξειδίκευσης Έλληνες εργαζόμενοι εκεί. Αυτά πρέπει να λέμε στην έκθεση, όχι να μιλάμε για ζητήματα νομιμοποίησης. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Λάγκεν και να δώσουμε τώρα το λόγο σε έναν συνάδελφο από την Γερμανική Βουλή, στον κύριο Κυρία Πρόεδρε. Θα παραθέσω τα λόγια προηγούμενου Προέδρου της Γερμανίας. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάθε φορά που δείχνουμε με το δάχτυλο κάποιον, τρία δάχτυλα δείχνουν προς τη δικιά μας μεριά. Και θα ήθελα μια πιο διαφοροποιημένη συζήτηση. Τα κράτη βρέθηκαν στην κρίση για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετική ένταση. Ο προλαλής σας προσπάθησε να το θέσει αυτό κομματικά. Αυτό δεν εξηγεί όμως την κατάσταση στην Ιρλανδία. Κύριε Λάνιε, θυμάμαι πριν 10-15 χρόνια που η Ιρλανδία αναφερόταν ως μοντέλο στην ε, Ευρώπη ως οικονομία το μέλλον θεωρήθηκε τότε ότι ε, ανήκει στις υπηρεσίες και μάλιστα στις ε, χρηματοοικονομικές. Ε, ξέρουμε τώρα ότι η φούσκα αυτή έσκασε, ότι πρέπει να διασωθούν οι τράπεζες και ότι η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Ιρλανδία. Ο Ιρλανδός συνάδελφος αναφέρθηκε στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Κάτι που στην Γερμανία αποτελεί πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν σας παρακαλώ να συζητάμε με πιο πολλές αποχρώσεις. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν αρκετές προκαταλήψεις και ε, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Πριν 10-15 χρόνια ε, ε, θεωρούμασταν ο ασθενή της Ευρώπης, ενώ σήμερα η παραγωγή μας θεωρείται πλεονέκτημα. Η μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 2000 Ε, δεν είχε να κάνει μόνο με τη λιτότητα. Χρειάζεται χρόνο ώστε οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις να παρουσιάσουν αποτελέσματα. Πιστεύω ότι ναι, η Τρόικα σε κάποια σημεία υπερέβαλε. Ε, δεν αρκεί εξυγίανση όταν χρειαζόμαστε και ανάπτυξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ε, δεν είναι υπεύθυνε οι εθνικέ κυβερνήσει και τα εθνικά κοινοβούλια. Χρειαζόμαστε την σωστή ισορροπία στη συζήτηση. Η υπόλωση δεν θα μα βοηθήσει τελικά. Και διότι ε, αυτή μάλλον βλάπτει την, ε, τη θέση της Ευρώπης σε όλα τα κράτη-μέλη. Συνάδελφο Σάουρα, Πέντρο Σάουρα από την Ισπανική Γερουσία. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ είμαι υπέρ μιας πιο συνεργατικής εντός εισαγωγικών συζήτησης. Μην θεωρούμε ότι διασώσαμε το ευρώ με τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την οικονομική ανάπτυξη. Καταρχάς, διότι σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές μας περιμένει μία μακρά περίοδος ε, στασιμότητας από οικονομική σκοπιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Με ανησυχεί επίσης και το γεγονός ότι υποφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλές οικογένειες και ε, στην πραγματικότητα πλήττεται και το μέλλον του ευρωπαϊκού προγράμματος. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τα σφάλματα του παρελθόντος, ε, τόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά όσο και τα εθνικά κοινοβούλια. Η κατάσταση στη χώρα μου δεν έχει σταθεροποιηθεί, εξακολουθούν να μειώνονται οι πιστώσεις, ε, η ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται, καταργούνται θέσεις εργασίας, καταστρέφονται επιχειρήσεις και η οικονομική ανάπτυξη, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν φτάνει στις περισσότερες οικογένειες. Δεν σταθεροποιείται το δημόσιο έλλειμμα και δεν σταθεροποιείται το δημόσιο χρέος. Να σας δώσω ένα αριθμητικό στοιχείο. Τα τελευταία δύο χρόνια το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 22,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και οδεύουμε ολοταχώ προς το 100% του ΑΕΠ σε πολύ λίγους μήνες. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε, όπως σα είπα και προηγουμένω να αντλήσουμε διδάγματα από τα σφάλματα του παρελθόντος. Ναι, ενεργή οικονομική πολιτική, αλλά μία δημοσιονομική πολιτική πρωτίστω στι χωρε που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο. Μία ε, πολιτική σταθεροτητα ε, ναι, αλλά με... Ε, σοφροσύνη και με αξιοπιστία. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν θα πρέπει και αυτές να ξεχνούν σε ποια χώρα γίνονται. Δεν θα πρέπει να ξεχνούν ποιος είναι ο οικονομικός κύκλος. Δεν θα πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι θα πρέπει να γίνει ταχύτατα διαχωρισμός ε, μεταξύ ε, του κινδύνου του δημοσίου χρέους και του τραπεζικού κινδύνου. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ανισότητα όχι μόνο ως διοντολογικός και ως ηθικός παράγων, αλλά και ως σταθεροποιητικός παράγων. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία βορανότου, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ χωρών ε, δωρητών και χωρών που είναι υπόχρεες στις πολύπες. Ευχαριστώ. Αδελφός Φένες από το Κοινοβούλιο της Μάλτας. Thank Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι έχοντας ακούσει αρκετούς ομιλητές θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι ενώ είναι σημαντικό να μιλάμε για τη δημοκρατική νομιμότητα της Τρόικας, πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε και για την ευθύνη. Είναι άδικο να προσπαθούμε να κατηγορήσουμε για τα προβλήματα της Ευρώπης, την ανεργία, ε, την ε, φτώχεια, ε, τα δύσκολα προγράμματα, να τα φορτώνουμε όλα στην Τρόικα και τις αποφάσεις της. Γιατί στην πραγματικότητα τα προβλήματα δημιουργήθηκαν από τις νόμιμα εκλεγμένες κυβερνήσεις, τα μέλη του Κοινοβουλίου, που την περίοδο των παχιών αγελάδων αποφάσισαν να παράσχουν υπερβολικά προνόμια στους, ε, ε, στο λαό τους, ε, μεγάλες, ε, μεγάλα επιδόματα, μεγάλες συντάξεις που δημιούργησαν προβλήματα και την ώρα της κρίσης η Ευρώπη λύγησε. Και γι' αυτό τώρα συζητάμε θέματα αλληλεγγύης. Είναι λοιπόν πολύ άδικο να λέμε στον χειρουργό ότι εσύ φταίς που πονάει ο ασθενής την ώρα που κάνει την εγχείρηση και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε πώς μπορεί η Τρόικα να λειτουργήσει με κοινοτικές μεθόδους όταν βυθίζεται το πλοίο. Την ώρα εκείνη χρειαζόμαστε τεχνοκράτες που θα μας δώσουν τεχνικές γνώμες και βοήθεια για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Να πω ακόμη ότι κάθε χώρα που μπήκε σε μνημόνιο αντιμετώπισε αποφάσεις της Τρόικας που έπρεπε όχι να εφαρμοστούν άμεσα αλλά να περάσουν από τα κοινοβούλια τα οποία διόρθωσαν τις, ε, ενδεχομένως τις αποφάσεις της Τρόικας για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από άλλα κράτη-μέλη και να στηριχθεί η οικονομία τους. Πρέπει λοιπόν να ε, έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση σχετικά με το που, ε, ποιον κατηγορούμε. Αυτές είναι ευθύνες κοινέ. Ο συνάδελφος Ρωσάτη από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων στον προηγούμενο ομιλητή γιατί με κάλυψε σχεδόν ολοσχερός. Δεν πρέπει να συγχέουμε τα τεχνικά ζητήματα με τα πολιτικά. Βεβαίω η Τρόικα δεν είναι δημοκρατικός θεσμός με την παραδοσιακή έννοια του όρου, είναι τεχνοκρατικό σώμα με καθήκον να κάνει μια αξιολόγηση αντικειμενική μιας κατάστασης και να προτείνει λύσεις. Και τα πολιτικά σώματα, οι δημοκρατικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια θα λαμβάνουν τις αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνέπειες και τις εναλλακτικέ. Δεν πρέπει να περιμένουμε από τα κοινοβούλια να συζητούν τα τεχνικά θέματα των προγραμμάτων προσαρμογής πρέπει να παίρνουν αποφάσεις αν θα συνεχίζουν τα προγράμματα προσαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τα υπέρ και τα κατά τους και θα αποφασίζουν θα τα υλοποιήσουν ή όχι. Οι εμπειρογνώμονες μπορεί και να ασφάλουν βέβαια. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπάρχει εμπειρία. Το Νομισματικό Ταμείο στις δραστηριότητες του σε διάφορες χώρες έκανε κατά το παρελθόν λάθη. Και ξέρουμε ότι οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές σε εποχές ύφεσης είναι μεγαλύτεροι από ό,τι τους είχαμε υπολογίσει πριν. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι η αντίληψη ότι η κοινοτική μέθοδος θα μας είχε επιτρέψει να αποφύγουμε το σφάλμα αυτό και θα είχαμε τότε καλύτερη κατανόηση της κατάστασης από τα πριν, δεν είναι ρεαλιστική. Δεν είναι καθόλου ρεαλιστική αυτή η άποψη. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Αντολίν Σάνσας Πισέτο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς να σας πω ότι εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι δύο συνεισυχητές θα καταλήξουν σε μια πολύ καλή έκθεση και ότι προκειμένου να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση, κατά την άποψή μου θα πρέπει να ενισχύσουμε το δημοκρατικό έλεγχο των κοινοβουλίων ε, και ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η Τρόικα αποτελεί τμήμα της ε, αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά η κρίση έχει τουλάχιστον τρία στάδια. Το ένα είναι η πρόληψη, στο οποίο κατά την άποψή μου υπήρξαν σφάλματα, διότι δεν υπήρχε οικονομικός έλεγχος και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και είναι προφανές ότι δεν υπήρχε οικονομικό συντονισμός, υπήρχε ένα έλλειμμα οικονομικής διακυβέρνησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν αξιολογήθηκε επίσης και καταλήλως στα εθνικά κοινοβούλια ο κίνδυνος ο οποίος μπορούσε να προκύψει. Και υπήρχαν χώρες οι οποίες χρεώθηκαν πάρα πολύ, αλλά μεγάλο τμήμα του χρέους έχει ως πιστωτές άλλες χώρες οι οποίες εμπιστεύτηκαν τις χώρες αυτές και προφανώς ε, τη στιγμή στην οποία προέκυψε η κρίση δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε και να αφήσουμε την ευθύνη μόνο σε μερικούς, διότι ήταν ε, ε, κοινή η ασυδοσία από όλες τις πλευρές. Και επομένως θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις ε, στην οικονομική διακυβέρνηση, στο συντονισμό και στην αντιμετώπιση των, των κινδύνων και ε, στο τμήμα της διαχείρισης της κρίσης. Εκεί είχαμε διακυβερνητική διακήρυξη και επομένω είναι ευπρόσδεξη αυτή η αντίδραση. Άλλο βέβαια είναι το γεγονός ότι στο μέλλον θα πρέπει να προέχει κάποια άλλη μέθοδος. Θα χρειαζόμαστε κάποια πιο αποτελεσματικά μέτρα. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε αποφάσεις ε, και κάποιος ε, να επιβάλλει προϋποθέσεις και να θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός σταθερότητας, πρέπει να τον διαθέτουμε, θα πρέπει να κινητοποιείται κατόπιν μιας ευρωπαϊκής προοπτικής και αυτό θα πρέπει να ενισχύσει το ρόλο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τα Εθνικά Κοινοβούλια, διότι αυτά το είναι ε, ε, που θα ελέγχουν τους εκπροσώπους τους ε, στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ελέγχει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, για την Τρόικα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το βασικό ρόλο των προγραμμάτων προσαρμογής, των μνημονίων. Αλλά τα μνημόνια είναι και προγράμματα σταθερότητας της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι γίνονται αντιληπτά απλώς προγράμματα προσαρμο... ως προγράμματα προσαρμογής των χωρών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα συνοδευτικό πρόγραμμα και θα πρέπει να υπάρχουν και συνοδευτικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ο ρόλος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να διασφαλίζει ότι η νομισματική πολιτική θα είναι προ όφελο των μνημονίων και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο κλήθηκε διότι ήταν ο μόνο διεθνή οργανισμό που μπορούσε να ε, διασφαλίσει πολυμερή ε, βοήθεια. Και θα πρέπει στο μέλλον να έχει διαφορετικό ρόλο. Θα πρέπει να διαφυλάξει την ε, διεθνή οικονομική σταθερότητα. Και δεν μπορούμε να ζητούμε από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να μην διαδραματίζει το ρόλο του. Και υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό η ανάκαμψη. Πρόληψη, διαχείριση και ανάκαμψη. Και νομίζω ότι εδώ τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να σκεφτούν λίγο. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις υπάρχουσες ανισορροπίες δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε το ίδιο. Θα πρέπει όλοι με κάποιο τρόπο να συνεισφέρουμε στην ανάκαμψη. Στο λόγο ο κ. Γεργέρη από την Ιταλική Γερουσία Επιτροπής Uh, e- θα ήθελα να μιλήσω για την οικονομική αποτελεσματικότητα του προγράμματος της Τρόικα, διότι όταν υπάρχει έλλειψη δημοκρατική νομιμο... δημοκρατικής νομιμοποίησης και συμφωνώ με τους ομιλητές στο βήμα, εάν δούμε την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα δούμε ότι είναι ανάμεικτα υπάρχουν ε, τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά αυτά ε, διαφέρουν από την πραγματική οικονομία. Είδαμε ότι η ανεργία έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ότι η ύφεση είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι περιμέναμε. Αυτό δεν, σημαίνει, δεν συμβαίνει λόγω έλλειψης οικονομικής εξυγίανσης, διότι ξέρουμε ότι όλα όλες οι χώρες ε, των προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας έχουν κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι είχαν προγραμματιστεί στο μέτωπο αυτό. Το πρόβλημα ήταν η κατάρρευση του ΑΕΠ. που έριξε τη χώρα σε μια παγίδα ύφεση και δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. Το ερώτημα είναι, η Τρόικα θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Η απάντησή μου είναι ναι και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο βασικά λάθη. Αλλιώς το μέλλον δεν θα είναι πιο φωτεινό. Τα δύο λάθη, όπως είπαν και άλλοι, ήταν ότι καταρχάς η Τρόικα δεν υπολόγισε σωστά τις συνέπειες ε, της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των περικοπών. Υποτίμησε την, ε, τη μείωση, την αύξηση της ανεργίας και αυτή είναι η λεγόμενη ιστορία των πολλαπλασιαστών. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πολλαπλασιαστές δεν είναι σταθεροί όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλάζουν κατά τη διάρκεια του κύκλου. Ε, αυτό θα ήταν μια πολύ σημαντική βελτίωση. Δεύτερο λάθος, η Τρόικα δεν πρόσεξε αρκετά τις συνέπειες από τη μία χώρα στην άλλη. Εξέτασε κάθε χώρα μεμονωμένα. Δεν εξέτασε τα συστημικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι το φάρμακο που δόθηκε έχει αρνητικές συνέπειες. Το πρόβλημα είναι ότι το φάρμακο δόθηκε σε λάθος δόσεις. Χρησιμοποιήθηκαν λάθος μέθοδοι διότι αλλιώς στο μέλλον θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό θα ήταν μεγάλο λάθος. από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Euh, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου κύριε Πρόεδρε να σας πω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε όλα. Επικροτώ το γεγονός ότι μπορέσαμε να διασώσουμε το ευρώ, ότι μπορέσαμε να βοηθήσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ακόμα και αν ε, υπάρχουν κάποιες πτυχές και κάποια μέτρα τα οποία έλαβαν οι Τρόικα, τα οποία δεν επικροτούμε. Χρειάστηκε όμως να εφαρμοστούν κάποιες λύσεις κατεπηγόντως και νομίζω ότι δράσαμε στη διάρκεια εκείνης της επίγουσας κατάστασης και τώρα καλώς κάνουμε και σκεφτόμαστε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, ε, τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, τι θα πρέπει να γίνεται, αλλά θα πρέπει να πω ότι υπάρχει κοινή ευθύνη μεταξύ των χωρών που διέπραξαν σφάλματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν κατάφερε να τους προλάβει και που δεν κατάφερε να διαβλέψει ότι ε, θα διαπραχθούν σφάλματα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτα πρέπει να διορθωθεί αυτό. Θα πρέπει να διορθωθεί το γεγονός ότι... Ε, ο κόδωνας του κινδύνου δεν έκρουσε και επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις εξουσίες της Eurostat και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορεί να προβλέπει απευθείας τι μπορεί να συμβεί και επίσης θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να διστάζουμε. Υπάρχει το άρθρο 13 της συνθήκης. Εγώ συμμετείχα στην πρωτοβουλία για αυτό το άρθρο 13 και όλοι τώρα λέμε ότι το Εθνικά Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργάζονται. Θεωρώ όμω ότι είναι πονδύδιστο το γεγονό ότι στην ε, διάσκεψη του Βίλνιου δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι δεν μου φαίνεται καλή λύση να υπάρχει ένα κοινοτικό ε, νομισματικό ταμείο. Θα αποφασίσει βέβαια στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και τι ευθύνη ελέγχου έχουν τα κοινοβούλια για τις δανειοδοτήσεις που προσφέρονται στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και επίσης θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα προφανώς και τα αντιλαϊκά κινήματα ε, τον ευρωσκεπτοκισμό, ο οποίος δημιουργείται και στις χώρες οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση, αλλά και στις χώρες δωρητές. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και στις δύο ομάδες χωρών. Και τέλος ε, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να βρούμε τη δέουσα ισορροπία μεταξύ ε, υποστήριξης της ανάπτυξης και κατάλληλου ελέγχου των ε, δημοσίων λογαριασμών και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το χρέος του ιδιωτικού τομέα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπογράμμισε ότι το βασικό στοιχείο της ανάπτυξης είναι να προσέξουμε πόσο σημαντικό είναι το χρέος στο ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Περβάνς Μπερές, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συγητές, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Λάγκεν. Δυστυχώς έφυγε βέβαια. Ο κύριος Βέρνερ Λάγκεν είναι εδώ. Εντάξει, καλύτερα ακόμα. Επικρίνατε, κύριε Θέρκας, ε, ε, τα όσα συνέβησαν στην Ισπανία, αλλά δεν ήταν μόνο στην Ισπανία. Και θα ήθελα να πω ότι πριν από την κρίση η Ισπανία ήταν στους καλούς μαθητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πληρούσε τα λεγόμενα κριτήρια του Μάστριχτ κύριε Λάμπερτ, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτησή μας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο δημοκρατικός χώρος σε παγκόσμια κλίμακα βάσει των ε, ε, ε, μελετών, ότι αυτό θα πρέπει να μας αρκεί και ότι δεν θα πρέπει να δίνουμε χρηματοδότηση χωρίς να επιβεβαιώνουμε και τα προγράμματα και επειδή έγινε μια επικύρωση του προγράμματος στο Eurogroup αυτό δεν αποτελεί δημοκρατική νομιμοποίηση. Όσον αφορά την Τρόικα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε δύο διαστάσει που νομίζω ότι έχουμε υποτιμήσει στη σημερινή συζήτηση. Οι χώρε οι οποίες ε, ε, κάνουν διαστροτική ε, μεταρρύθμιση σε καλέ συνθήκε, είναι χώρε τις οποίε ο κοινωνικό διάλογο βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Όπου παρεμβαίνει η Τρόικα δεν ασχολείται καθόλου με τον κοινωνικό διάλογο και αυτό το επανέλαβε και η Διεθνή Οργάνωση Εργασία και το Συμβούλιο τη Ευρώπη στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ό,τι συμβαίνει εκεί δεν θα μπορούσε να συμβεί και αλλού. Όλοι οι Ευρωπαίοι αναφέρονται στο benchmark, στο ε, μαθαίνω ε, μέσω εφαρμογής πραγμάτων και αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Κάποιες χώρες οι οποίες καταφέραν να ε, επιτύχουν μετά την παρέμβαση της ε, Τρόικας δεν θα πρέπει να τις ε, εξετάζουμε μόνο με βάση συγκεκριμένου παράγοντε, θα πρέπει να λαμβάνουμε επίση υπόψη και τη μετανάστευση. Στην περίπτωση της Λετωνίας, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι είναι μια χώρα η οποία διέφυγε τον κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού, οι νέοι, μετανάστευσαν και ουσιαστικά θα δημιουργήσουν τα προβλήματα του αύριο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπερέ. Το λόγο έχει ο κύριος Καριέλο από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή όλων στα όσα μας ενδιαφέρει στη σημερινή συζήτηση, δηλαδή τη δημοκρατική νομιμοποίηση των ε, μνημονίων. Εγώ θεωρώ ότι αντί να αναφερόμαστε σε δημοκρατική νομιμοποίηση, θα έπρεπε να αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο είναι εντελώς παράνομο, το οποίο το περάσαμε ε, μέσω ε, δημοκρατικού τρόπου και αναφερόμαι στο Fiscal Compact, στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ε, αναφέρθηκε σε, μία, ε, σε έναν ισοσκελισμό των προπολογισμών συμπεριλαμβανομένων και των όσων περιλαμβάνονται στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ποιος είναι αυτός που αποφασίζει αν δεν αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Εάν μπορέσαμε να παρακάμψουμε μία συνθήκη η οποία ενώνει και επί της οποίας θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος κάποιων χωρών με το μακρύ χέρι της Τρόικας, αν αυτό δεν υποσκάπτει τη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αυτό δεν δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο, διότι εδώ όλοι συμφωνούμε νομίζω και όλοι είπαν ότι οι ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο στις διάφορες ε, χώρες μέλη είναι προφανείς. Υπάρχει συνεχής ε, ανεργία, αυξανόμενη, υπάρχει δυσκολία πρόσβασης σε πιστώσεις και χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις και υπάρχει ένα φαινόμενο ύφεση σε σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν αυτές είναι οι συνόπιες και αν η πράξη είναι παράνομη, διότι το πρωτόκολλο υπαριθμών 12 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιβαίνει σαφώς το άρθρο 3 του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Κυρίες και κύριοι λοιπόν, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η δημοκρατική νομοποίηση αυτής της πράξης. Και θα πρέπει να υπάρξει και η ρήτρα της επαναχώρησης, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουν όλες οι χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κ. Χρυσόγελος. Ε, νομίζω ότι ένα σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που ζητάει το Κοινοβούλιο, δηλαδή ότι κάθε πολιτική, δημοσιονομ... κάθε πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής πρέπει να αξιολογείται και να διορθώνονται τα λάθη και να αλλάζει πολιτική αν αποτυγχάνει στόχους ε, και αυτό πρέπει να γίνεται σε διάλογο με την κοινωνία και τους πολίτες στην κοινωνία των πολιτών και όχι μόνο με τις κυβερνήσεις και το κοινοβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οποιαδήποτε πολιτική ε, όταν ασκείται πρέπει να αξιολογείται, να κοιτάμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και να διορθώνουμε και να βλέπουμε πέρα από την στιγμή που ήταν η κρίση μετά από 5-6 χρόνια ποιες είναι οι επιπτώσεις και στους άλλους τομείς γιατί δεν μπορεί να μην βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην κοινωνία και στο περιβάλλον στην κοινωνική συνοχή, στην απασχόληση στην ίδια την παραγωγική βάση της χώρας. Επομένως αν κάποιο μπορεί να δικαιολογήσει λάθη τη στιγμή τη κορύφωση κρίση, δεν μπορεί μετά από 5-6 χρόνια να δικαιολογεί αυτέ τι πολιτικέ, όταν βλέπουμε ότι έχει αστοχήσει πλήρω. Ξεκίνησε η πολιτική αυτή να ε, προσπαθεί να μειώσει το έλλειμμα, Όμω, σήμερα έχουμε τεράστιο χρέο, έχουμε τεράστια ενεργεία, 28% και πάνω από το 60% για τους νέους, έχουμε ύφεση 35%, έχουμε 30% των ανθρώπων ανασφάλιστοι σήμερα σε μια χώρα ευρωπαϊκή και πάνω από 1,5 εκατομμύριο χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Ακόμα και αν πετύχουμε δημοσιονομικούς στόχους που δεν τους έχουμε πετύχει, αυτή η πολιτική φαίνεται έχει αποτύχει. Υπάρχουν λοιπόν μερικά προβλήματα. Πρώτον, η μέθοδος, δηλαδή η Τρόικα, ήταν εκτός κοινοτική μεθόδου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει τους πρώτους έξι μήνες τον πρώτο χρόνο ήταν μια κατάσταση κρίσης είχαμε προβλήματα δημοσιονομικά είχαμε προβλήματα αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης αλλά σήμερα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει εκτός κοινοτικής μεθόδου. άρα δεν μπορεί να νομοποιείται μια, ένας θεσμός που λειτουργεί εκτός κοινοτικής μεθόδου. το δεύτερο είναι ότι και οι πολιτικές απέτυχαν όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος αλλά σήμερα διαπιστώνουμε ότι και οι προποθέσει που χρησιμοποιήθηκαν όπως ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής ή υποτιθέμενες επιπτώσεις είναι πλήρως άστοχες. Άρα λοιπόν πρέπει νομίζω να τελειώσει η Τρόικα, πρέπει να πάρουμε υπόψη όλη αυτή την εμπειρία, να δημιουργηθούν οι θεσμοί εκείνοι που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις αλλά θα προλαμβάνουν και τις κρίσεις και κυρίως τώρα πρέπει να επανέλθουν αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται ώστε να είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή στρατηγική και τις άλλες πολιτικές το Ευρώπη 2020, την οικολογική καινοτομία, το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή μετά από 5-6 χρόνια δεν μπορεί πλέον να λέμε ότι δεν ξέρουμε ότι μπορεί να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Και το λόγο έχει η κυρία Μορτάγκουα από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας, Μαριάννα Μορτάγκουα. Um, Ευχαριστώ κυρία, κύριε, ε, κύριε Πρόεδρε. Έγινε αναφορά και στη χώρα μου και τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας της, παραγωγή, περιφερική θέση της χώρας, περιφερειακή θέση. Για πολύ καιρό ήταν ε, χαμηλότερο το έλλειμμα το, ε, από το εκείνο της Γερμανίας, ε, κάτω από 3%. Είχε επίσης χαμηλά επίπεδα ανεργίας. Όμως η χρηματοπιστωτική κρίση τα άλλαξε αυτά τα δεδομένα και στην Πορτογαλία και αλλού. Αυξήθηκε από 12% η ανεργία το 2000, αυξήθηκε από το 12%, αυξήθηκε το χρέος, ε, υπάρχει πρόβλημα ε, με χρηματοδότηση. Θα έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την ε, Τρόικα που επέβαλε λιτότητα δεν υπήρχε ε, πλήρης ε, συμφωνία από το Κοινοβούλιο στα μέτρα αυτά. Επίσης ε, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα με τα προγράμματα αυτά μετά λόγω της νομιμότητας. Ένα πρόγραμμα προσαρμογής όπως το πρωτογαλλικό αντίκειται και στο σύνταγμα αυτών των χωρών. Υπάρχει και ένα τεχνικό ζήτημα. Το μνημόνιο της Τρόικας για την Πορτογαλία στηρίζεται σε εικονικούς δείκτες. Οι, προγνώση, οι προβλέψεις έπρεπε να αλλάζουν ε, πολύ βραχυπρόθεσμα γιατί δεν ίσχυαν, αποδεικνυόταν ότι δεν ε, ίσχυαν. Και τα αποτελέσματα των μνημονίων. Κανένα ε, πρόγραμμα δεν επηρέασε το έλλειμμα. Το έλλειμμα είναι ε, περίπου όπως ήταν και το χρέος αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Απότομα. Το ΑΕΠ αυξήθηκε λίγο, αλλά οι εσωτερικές ανισότητες οξύνθηκαν. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι ε, έγιναν φτωχότεροι, αυξήθηκαν οι εκατομμυριούχοι και τώρα έχουμε ε, προβλήματα που δεν τα είχαμε ε, δει ε, μετά το τέλος της επικιοκρατίας. Περίπου μισό εκατομμύριο είναι οι άνεργοι και το ενεργός πληθυσμός είναι 5 εκατομμύρια. Είναι ακραίες αυτές οι καταστάσεις και είναι και περίεργο που αναφέρεται σε αυτό το κοινοβούλιο ότι τα μνημόνια ήταν αποτελεσματικά. Για τους φτωχούς δεν ήταν. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να κινηθούμε υπέρ των πολιτών. Η κυρία Φερέιρα. Um, Ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή. Πρέπει να πω καταρχήν ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε ότι η δημιουργία κοινού νομίσματος απαιτεί κάτι παραπάνω από σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Γιατί ε, δεν υπάρχει εγγενής μηχανισμός σύγκλησης, αλλά απόκλησης. Αυτό πρέπει να προλάβουμε για να τελειώσει η κρίση. Η κρίση έλαβε χώρα και εμείς δεν είχαμε επαρκείς μηχανισμούς επίλυσης. Πρέπει να τελειώσει αυτή η περίοδος ε, με μηχανισμούς ενσωματωμένους στο ενίο νόμισμα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλω να περάσω. Βεβαίως χρειάζεται και μια αποτελεσματική τραπεζική ένωση, όχι οποιαδήποτε τραπεζική ένωση. Και πρέπει να δούμε και τι προϋπολογισμό έχουμε στη διάθεσή μας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε μια νέα κρίση. Ο ε, ESM δεν αρκεί. Πρέπει να δούμε αν η Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσης αν σε δια... Ε, αντιπαράθεση με την ε, Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, την οικονομία όταν δεν υπάρχει πληθωρισμός και πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα της έρευνας ε, της Επιτροπής μετά από πιέσεις του Κοινοβουλίου. Ε, να δούμε πώς μπορεί να σταθεροποιηθεί το δημόσιο χρέος, αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός και μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο κοινό σύστημα εγγυήσεων όταν αναγκαζόμαστε να ακολουθούμε προγράμματα προσαρμογής που, που φορτώνουν βάρος, ε, βάρη υπερβολικά στο, στους λαούς μας. Ε, όταν δηλαδή υπάρχει ε, πρόβλημα στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και όταν αυξάνεται η φτώχεια. να δούμε και τα τεχνικά ζητήματα των συστάσεων. Κοινωνικό κόστος, αυξανόμενο κόστος, τελειώνω. Έχουμε όμως ύφεση, ε, μειώσαμε την ανάπτυξη, μειώθηκε η ανάπτυξη και ένα άλλο πρόβλημα είναι οι ιδιωτικοποίησεις που επευλήθησαν σε αυτές τις χώρες ε, στον τομέα τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικής ενέργειας, στον τραπεζικό τομέα, τον ασφαλιστικό τομέα, ταχυδρομεία. Αυτά θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όπως και οι στρατηγικές επενδύσεις. Χρειάζονται λοιπόν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συγγνώμη που ξεπέρασα το χρόνο. Το λόγο έχει ο κύριος από το Κροατικό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την οργάνωση αυτής της διάσκεψης. Θα μιλήσω κροατικά. Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι για να πετύχουμε προ πρόοδο και να πετύχουμε μακροοικονομική σταθερότητα, όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη εφαρμογή των μέτρων. Γι' αυτό είναι μεγάλης σημασίας να έχουμε καλή επικοινωνία, καλή επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τα οικονομικά μέτρα προσαρμογής και που στόχο έχουν ε, την εξασφάλιση της ανάπτυξης και της απασχόλησης δεν μπορούν να πετύχουν χωρίς, ε, εάν δεν λάβουμε υπόψη, την πραγματική οικονομία. Συζητάμε λοιπόν τη δημοσιονομική εξυγίανση, τις ε, μακροοικονομικές προκλήσεις, την δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν έχουμε συζητήσει όμως το θέμα της αποτελεσματικότητας, ούτε έχουμε λάβει απαντήσεις όσον αφορά τους τρόπους διασφάλισης της αποτελεσματικότητας, κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε το μέλλον. Για να είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες μας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, την ε, πραγματική οικονομία. Να ρωτιέμαι αν έχουμε ξεχάσει τα πάντα περί κοινοπαξιών ε, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Ίσως ε, επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στην Τραπεζική Ένωση. Η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις. Και τίθεται το θέμα εάν έχουμε επαρκή αριθμό μέτρων για να διασφαλίσουμε την μελλοντική ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τις Εθνικές Τράπεζες για να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στην μελέτη ανεξάρτητης ανάπτυξης 2013-2014 όπου διαπιστώνεται ότι δεν ήταν επιτυχημένα τα μέτρα. Γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ε, άλλωστε εκπροσωπούμε τους πολίτες μας ε, και τα μέτρα λιτότητας έχουν πολλά θύματα. Ανέργους, ανθρώπους με επισφαλείς θέσεις εργασίας και φυσικά υπονομεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουμε λοιπόν το πρόβλημα της φτώχειας. Επίσης βλέπουμε να υπάρχει μυσαλλοδοξία και εξτρεμισμός. Η Ήπειρός μας νόμιζε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, έχουμε κρυζώσει τα φαινόμενα αυτά. Όλα αυτά έχουν ε, τεράστιες συνέπειες για τους πολίτες μας. Επίσης ε, βλέπουμε μία προηγουμένου διαφυγή εγκεφάλων, διαφυγή των ικανών ανθρώπων δηλαδή από την Ευρώπη και η νέα γενιά αναζητά ένα καλύτερο μέλλον, ακόμα και μακριά από την Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να παραθέσω έναν από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους, τον Κέινς, που είπε ότι για να μειωθεί η ανεργία ε, της μεγάλης κρίσης ε, του 1930 ήταν απαραίτητο όχι μόνο να ληφθούν μέτρα λιτότητας, οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να προσέξουν την ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι πολλοί είναι αναγκασμένοι να αναλαμβάνουν επισφαλείς θέσεις κάτι που δεν οδηγεί όμως στην οικονομική ανάπτυξη. Τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της γραφειοκρατίας. Επίσης, Ήρθε η ώρα να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες μας. Η οικονομία της Ευρώπης μπορεί να αποκατασταθεί. Με κυβερνητικά προγράμματα και με προγράμματα του ιδιωτικού τομέα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει λύση η οποία να παράσχει ε, καλύτερο βιωτικό επίπεδο στους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. και παρότι προφανώς υπάρχουν ε, διεστάμενες απόψεις, δεν θα μπορούσε άλλωστε να συμβαίνει κάτι διαφορετικό καθότι υπάρχει και πολλή φιλολογία πάνω στο θέμα αυτό και όχι μόνο ε, ε, οικονομικά κείμενα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα του τι εννοούμε και πώς ε, ορίζουμε την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση. Υπάρχει πάντως νομίζω συνένεση πάνω σε δύο θέματα. Καταρχάς σε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκπονήσει την έκθεση αυτή. Είναι μια σημαντική απόφαση διότι προκάλεσε μια δημόσια συζήτηση πάνω στη διαδικασία, πάνω στο ρόλο και τις δραστηριότητες της, Τρόικα, Τρόικας. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν ότι λαμβάνονται αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών, κάτι που υπονομεύει την ε, ανάγκη για το αίσθημα οικειοποίησης. Και επίσης, σημαντικό Ποιοι είναι η ποιότητα της συζήτησης που μπορούμε να έχουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το συμπέρασμα αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το υπερασπιστούν και οι εθνικοί βουλευτέ και οι ευρωβουλευτές. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συμπρόεδρό μου και αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Γιάννη Τραγάκη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ομιλητές, τον Όρμπερτ Λάμερτ, πρόεδρο του Bundestag, τον Ντόμινικ Χάνιγκαν, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου και φυσικά τους δύο συνεισηγητές μας, τον Ότμαρ Κάρας και τον Λίεμ Γκότς. Και να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις παρεμβάσεις σας. Ε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δεμερτζόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής ε, Οικονομικών Θεμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να με βοηθήσει να συμπροεδρεύσουμε στο κομμάτι αυτό της συνεδρίασης.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 Okay. So we to... Uh, Προχωρούμε στην επόμενη ολομέλεια προώθηση της ε, ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη με τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να καλωσορίσω ένα πρώην συνάδελφο και φίλο, τον κύριο Έντουαρτ Σικλούνα, ο οποίος τώρα είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έντουαρντ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως ακούσατε, σιγά σιγά αυξάνεται η αυτοπεποίθηση ότι η Ευρώπη ε, ξέφυγε από την κρίση του χρέους. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη πόρο απέχει ακόμα από πλήρη ανάκαμψη. Αυτό νομίζω κατέστη σαφές και από την προηγούμενη συζήτηση. Και ακόμα είμαστε αντιμέτωποι με αρκετά θεμελιώδεις προκλήσεις. Μία από αυτές ε, είναι η συνεχιζόμενη και επίμονη στασιμότητα στην επενδυτική δραστηριότητα. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επιτάχυνε την κατάρρευση των επενδύσεων στην Ευρώπη. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, κατά 20% κάτω από το ανώτατο επίπεδο που είχαν το 2008, κυρίως λόγω της μείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Στις ε, πλέον πληγήσεις ε, χώρες της Ευρώπης οι επενδύσεις έπεσαν κάτω από 40% και ακόμη δεν υπάρχουν πιστικά σημάδια αναστροφής της κατάστασης. Η παρατεταμένη επενδυτική κρίση περιορίζει την ανάπτυξη στην Ευρώπη και σε σχέση με το ΑΕΠ και την απασχόληση και πόσο μάλλον σημαίνει μείωση της παραγωγής για χρόνια σύμφωνα με κάποιες ε, προβλέψεις, η μείωση των επενδύσεων στην Ευρώπη από το 2008 μέχρι το 2012 θα στοιχεί στην Ήπειρο 540 δις ευρώ σε ε, απώλεια απόδοσης μέχρι το 2020. Αυξάνεται το νούμερο αυτό και θα συνεχίσει να αυξάνεται στο βαθμό που θα είναι ε, μειωμένες οι επενδύσεις. Το ίδιο ανησυχητικό είναι ε, το γεγονός της επίμονης υψηλής ανεργίας σε πολλές νότιο-ευρωπαϊκές χώρες που διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει διαρθρωτικό το πρόβλημα και μαζί με το πρόβλημα το δημογραφικό θα, μειωθεί πάλι η, ε, θα μειωθούν οι εκροές και η παραγωγή στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δουλεύει σκληρά για να καταλάβει καλύτερα το, την κρίση και να ε, έχει καλή απόκριση. Οι συνάδελφοί μου στην ΕΚΟΡ όταν ήμουν εδώ Ευρωβουλευτής πιέζαμε για να υπάρξει αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πάνω σε αυτό το θέμα. Στο, στην καρδιά της κρίσης των επενδύσεων στην Ευρώπη βρίσκονται κάποιες διαρθρωτικές ανισορροπίες. Όπως γνωρίζουμε όλοι, κάποιες χώρες ε, είχαν μία επέκταση του δανεισμού, αύξηση του δανεισμού πριν από την κρίση και από εγχώριες και από ξένες πηγές και ο, αυξημένος δανεισμός οδήγησε σε αυξημένη κατανάλωση και υπερεπενδύσεις σε τομείς όπως ο, το, ο τομέας των ακινήτων. Εν μέρη τώρα βλέπουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις από αυτές τις υπερβολικές επενδύσεις. Μία επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη θα απαιτήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ούτως ώστε να πάνε οι πόροι σε πιο αποδοτικούς παραγωγικούς τομείς. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια τράπεζα ε, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μπορεί να στοχεύσει παρεμβάσεις ε, πέρα από τις συνολικές παρεμβάσεις για να προωθήσει τις επενδύσεις. Με τη βοήθεια της Τράπεζας Επενδύσεων μπορούμε να απαλείψουμε τα εμπόδια για την ανακατανομή των πόρων. Όχι μόνο για τις πλέον πληγήσεις χώρες αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η στόχευση των επενδύσεων είναι τόσο σημαντική. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, ένα πράγμα που μάθαμε είναι ότι ο ιδιωτικό τομέα συνολικά δεν περιορίζεται από έλλειψη χρηματοδότησης. Ε, κατά μέσον όρο, η μη χρηματο, τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βαρύνονται από, από χρέος. Μάλιστα, αύξησαν τις αποταμιεύσεις τους και έχουν γίνει καθαροί δανειοδότες, κυρίως στις κυβερνήσεις. Ε, αντιμέτωποι με ε, αβεβαιότητες σχετικά με την παγκόσμια οικονομία και τις προοπτικές για την Ευρωζώνη, οι ε, διοικητές κατάφεραν να υιοθετήσουν μια στάση του περιμένουμε να δούμε, αναβάλλοντας μεγάλες επενδύσεις μέχρι να δουν να μειώνεται η αβεβαιότητα που υπάρχει. Πάνω σε αυτή τη βάση είναι σαφές ε, ότι οι δεσμεύσεις ε, για την ακυριότητα της Ευρωζώνης ε, και οι νέες προτάσεις σχετικά με την Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να μειώσουν την αβεβαιότητα, να μετριάσουν τα χρηματοπιστωτικά εμπόδια που υπάρχουν, να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, αλλά όλα αυτά θα πάρουν χρόνο. Τώρα υπάρχει ανάγκη για καλά στοχευμένη δημόσια παρέμβαση όπου φαίνεται ότι υπάρχουν χρηματοδοτικοί περιορισμοί. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει τόσο κρίσιμο κέριο ρόλο κατά την κρίση. Ε, ένας υποτομέας ε, του ιδιωτικού τομέα που ε, επλήτεται και εξακολουθεί να πλήτεται από την κρίση είναι ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, ειδικότερα σε εκείνες τις χώρες που ε, πλήγησαν ε, ως επιτοπλίστων. Με τον κατακαιρματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών λόγω της κρίσης στην Ευρώπη, ο διασυνοριακός διδανισμός ε, περιορίστηκε στην Ευρώπη. Έτσι εξαρτώνται οι χώρες περισσότερο από την εγχώρια αποταμίευση και αυτό οδήγησε στην πανεμφάνιση σημαντικών εθνικών διαφορών στο κόστος δανεισμού ακόμα και μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτές οι αλλαγές έπληξαν σκληρά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφού εξαρτώνται ως επιτοπλίστων από τραπεζικό δανεισμό. Έτσι μετά την έναρξη της κρίσης το γεφύρωση του χρηματοπιστωτικού κενού για τις ΜΜΕ αποτέλεσε προτεραιότητα κύρια για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αφού αυτές οι ΜΜΕ παίζουν κρίσιμο ρόλο στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και ε, στις καινοτομίες. Ε, ο όμιλος της τράπεζάς μας εργάζεται για να λύσει τα χρηματοπιστωτικά προβλήματα με διάφορους τρόπους, ε, με στοχευμένο δανεισμό μέσα από χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές, ε, ούτως ώστε να ωφεληθούν ε, οι ΜΜΕ. Από τότε που άρχισε η κρίση, ο δανεισμός της ΜΜΕ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50% από 12 δις ευρώ στα 18,5 δις ευρώ το 2013. Παράλληλα, η ε, θηγατρική της Ευρωπαϊκής και Τράπεζας Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, υπέγραψε εγγύησεις για 2 δις ακόμη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε ε, εξετάσει πιλωτικά το μέσον Τζέρεμι για τις εγγυήσεις στη Μάλτα. Ε, ε, το δάνειο είχε αποτέλεσμα 10 μήνες πριν από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα Jeremy ε, βοήθησε πολλές επιχειρήσεις. Ε, η Τράπεζα της Μάλτας ε, μέσα από το Ταμείο Επενδύσεων εξέδωσε δεύτερη προκήρυξη ενδιαφέροντος για τον Αύγουστο 2013 στα πλαίσια του Jeremy για να βοηθήσει άλλες 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέρα από τις 530 που ωφελήθηκαν αρχικά. Ε, όμως ε, η ζήτηση για πιστώσεις αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και αυτό θα είναι πιο σημαντικό ακόμη για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, όμως ε, η τραπεζική χρηματοδότηση είναι ένα σκέλος των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Επειδή οι τράπεζες τώρα δυσκολεύονται να παίξουν το ρόλο τους και ε, να αναλάβουν ε, τον σχετικό κίνδυνο. Ε, οι ειδικέ γνώσεις της τράπεζάς μας επιτρέπει την υποστήριξη στην ανάπτυξη μέσων που κάνουν περισσότερο διαθέσιμη τη χρηματοδότηση από τις κεφαλαίες Πρωτοβουλίες για την βελτίωση της αντιμετώπισης των κινδύνων των ΜΜΕ βοηθούν στην προσέλκυση ε, νέων ευρωπαϊκών και διεθνών πηγών ε, χρηματοδότησης. Ε, όμως είναι λυπηρή αλήθεια ότι η ανεργία θα παραμείνει σοβαρό πρόβλημα ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που πέρασαν σε βαθιά ύφεση. Όταν ξαναρχίσει πάλι η οικονομική δραστηριότητα παρόλα αυτά θα υπάρχουν κάποιες ακαμψίες στην αγορά εργασίας σε χώρες όπου οι ε, επενδύσεις υποδομής ε, ε, έπεσαν κάτω από τις μακροπρόθεσμες τάσεις που είχαν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεχίζει να βοηθεί να μετριαστούν οι επιπτώσεις. Παράλληλα, οι διορθωτικές αλλαγές θα απαιτήσουν νέα εκπαίδευση, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που είχαν μεγάλο κατασκευαστικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μπορεί να στηρίξει ε, προγράμματα στην αγορά εργασίας ε, που θα έχουν ε, ένα ετήσιο ύψος 6 δις ευρώ, κυρίως για τις επενδύσεις, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση νέων. Η ανάπτυξη της στρατηγικής υποδομής παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δράση για τη βελτίωση του κλίματος, διευρωπαϊκά δίκτυα, ε, ο ρυθμός των επενδύσεων στις υποδομές έχει ζωτική σημασία ε, για την ανάκαμψη και την ε, μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επέκτηνε τις επενδύσεις στην υποδομή περισσότερο από 7,5 δις ευρώ από το 2012 μέχρι το 2013. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Ε, ομόλογα που συνδεδεμένα με προγράμματα και η ε, ε, συμβουλευτική από την τράπεζα ε, για καλύτερες δομές συμπράξεων ιδιωτικού δημοσίου τομέα μπορεί να βοηθήσουν να αυξηθούν οι επενδύσεις αποτελεσματικά προϊόντα όπως εγγυήσεις, δάνεια διαφόρων μορφών ε, θα υποστηρίζονται από τον μηχανισμό ε, διαρθρωμένης ε, χρηματοδότησης της τράπεζας. Ο ρόλος της τράπεζας θα συνεχίσει να είναι να προωθεί την σύγκληση μέσα από τη μόχλευση των ευρωπαϊκών πόρων, δρώντας ες καταλήτης βελτιώνοντας τις ε, ε, επενδύσεις ε, και κλείνοντας το επενδυτικό κενό. Και αυτή η κρίση όπως και άλλες άρχισε μια διαδικασία σημαντικών διαρθωτικών αλλαγών σε πολλούς κλάδους σημαντικούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συχνά συνδέεται με κοινωνικά προβλήματα. Έχει όμως και ε, κρυμμένες ευκαιρίες να λάβουν χώρα άλματα στην παραγωγικότητα μέσα από την καινοτομία. Και αυτό μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε ευημερία την Ευρώπη. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι βασικός περιορισμός για την καινοτομία, για καλύτερες τεχνολογίες και καλύτερες διαδικασίες που θα προκύψουν από την κρίση. Έτσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων άφησε τη οδανισμό στον τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης κατά περίπου 70%. Από 9,3 δις σε 15,6 δις ευρώ πέρσι. Παίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επιτυχών ε, εταιριών και κλάδων και βιομηχανιών της Ευρώπης του αύριο, ε, προωθώντας θετική οικονομική αλλαγή. Και για να πάω στα συμπεράσματα, η Ευρωπαϊκή και η Τράπεζα Επενδύσεων κάνει αυτό που αναμένεται από εκείνη. Ε, μετά την ε, αύξηση του κεφαλαίου ε, συνέβαλε σημαντικά στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση με αντικυκλικά μέτρα αναπτυξιακά. Το 2013 αύξησε το δανεισμό της κατά, περίπου, κατά περισσότερο από 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διατηρήσει τους ίδιους φιλόδοξους στόχους και φέτος και του χρόνου. Και είμαι βέβαιος ότι με αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και με καλά στοχευμένες στρατηγικές επένδυσεις και ανάπτυξης θα επανοικοδομήσουμε μια ακόμα ισχυρότερη Ευρώπη που θα προκύψει από την τωρινή κρίση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Um, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τις δικές σας παρεμβάσεις και να σας θυμίσω ότι μπορείτε να θέσετε και ερωτήσεις προς τον ομιλητή μας. Μπορείτε να συμπληρώσετε την ε, κάρτα που έχετε μπροστά σας και να μας τη στείλετε εδώ στο Προεδρείο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δερμερτσόπουλο που είναι πρόεδρος ε, της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να συντονίσει τη συνέχεια της συζήτησης. Ε, ξεκινάμε με τον κύριο Πάμπλο Ζάλμπα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ σχεδόν απόλυτα με τα όσα ακούσαμε από τον αγαπητού μας ε, φίλο τον κύριο Τσικλούνα. Νομίζω ότι περάσαμε από την κρίση χρέους Υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις οι οποίες μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση, αλλά θα πρέπει πλέον να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πολλό δε μάλλον σε ένα προεκλογικό πλαίσιο ε, όπου οι πολίτες θα μας ζητήσουν απτά αποτελέσματα. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε και βασικά στοιχεία. Καταρχάς τις μεταρρυθμίσεις. Οι χώρες οι οποίες είναι βυθισμένες στην διαδικασία της μεταρρύθμισης θα πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις και οι χώρες τις οποίες ε, σιγά σιγά βυθίζονται σε αυτή τη διαδικασία της μεταρρύθμισης θα πρέπει να δώσουν μια νέα μεγαλύτερη όθεση. Η άποψή μου όμως είναι ότι ακόμα μας περιμένει πάρα πολλή δουλειά θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε αντίστοιχες συνθήκες σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Είναι επονίδιστο το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται με βάση την τοποθεσία τους και όχι με βάση την οικονομική τους κατάσταση. Και παρά το γεγονός ότι αρχίζει να μειώνεται η χρηματοδότηση, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να βρούμε έναν τρόπο για να μπορέσει να χρηματοδοτούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να έχουμε αυτή την τόσο επιζητούμενη οικονομική ανάκαμψη. Οι πιστώσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ισπανία έπεσε κατά 11%. Ε, ακόμα και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Σίγουρα η Τραπεζική Ένωση θα μπορέσει να μας βοηθήσει, σίγουρα θα βοηθήσει να υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά αυτή η λύση είναι μεσομακροπρόθεσμη. Βραχυπρόθεσμα απαιτείται περαιτέρω δράση και κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν ιδιαίτερα στο ε, ε, πρόβλημα αυτό. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, η οποία θα πρέπει να είναι ακόμα πιο φιλόδοξη και να φροντίζει να φτάνει η χρηματοδότηση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ελπίζω στο επόμενο Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσει προ αυτή την κατεύθυνση. Και η δεύτερη είναι ο Ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μπορεί και πρέπει να κάνει κάτι περαιτέρω για το θέμα αυτό. Ε, δεν υπάρχει σαφής ε, ε, ε, διαβίβαση της νομισματικής πολιτικής και η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να δράσει προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κατάλληλη νομισματική πολιτική. Επιμένω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει και μπορεί να κάνει κάτι περαιτέρω επί του ζητήματος. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι ότι αν δεν φτάσει η πίστοση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύσκολα θα μπορέσουμε να έχουμε οικονομική ανάκαμψη η οποία θα είναι και εδρωμένη. Όλοι όσοι λοιπόν συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία θα πρέπει να δράσουμε και μάλιστα αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, ο κύριος ε, Πιέρ Αλέν Μιέ από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Oui, merci, le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωζώνη μόλις έκλεισε 2,5 χρόνια ύφεσης, ύφεση η οποία προέκυψε και ε, ε λόγω των προβλημάτων και γιατί προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και γιατί αναζητούμε μία ισορροπία μεταξύ του ελλείμματος και της ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές είναι αυξημένοι και υπάρχει ύφεση και αν όλες οι χώρες ταυτόχρονα επιβάλλουν πολιτικές λιτότητας, η μείωση του ελλείμματος δεν θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να δούμε τι συνέπειες θα υπάρξουν, διότι θα πρέπει ε, ναι με να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίαση αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα να αντισταθμίσει αυτή την ύφεση και να μπορέσει να επιβάλλει και κατάλληλες πολιτικές. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ τι γίνεται με την ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020 και τι γίνεται με το ε, Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλληλος ρυθμός μείωσης του διαρθρωτικού ελλείμματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσέξουμε ιδιαίτερα και τις πληθωριστικές τάσεις οι οποίες προκύπτουν από, το, ε, από την προσαρμογή των ισολογισμού και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και χθες. Και μια τρίτη παρατήρηση μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανακοδόμηση και η δημιουργία της ΕΚΑΧ ήταν μια πραγματικά εξαιρετική άγουσα προς την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση, την υπερθέρμανση του πλανήτη, τις κλιματικές αλλαγές και όλα αυτά θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, να έχουμε μια μεγαλύτερη ανάπτυξη και μια ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εχθές ε, ο πρόσωπος του ΩΣΑ μας υπενθύμισε ότι χρειαζόμαστε μεν διαρθρωτικές πολιτικές, αλλά είναι πιο αποτελεσματικές σε ένα κλίμα ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η Ευρώπη να ασχοληθεί με, με τη μακροοικονομία, αλλά ταυτόχρονα και με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος από την Πολωνική Βουλή, παρακαλώ. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλη μέρα συζητάμε θέματα που συνδέονται με την κρίση. Αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε κατά κάποιο τρόπο για τη δικαιοσύνη. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλες χώρες όπως είναι η Ινδία και η Βραζιλία, όπου η οικονομία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να σκεφτούν γιατί συμβαίνει αυτό. Έχουμε προγράμματα στήριξης, δίδουμε πιστώσεις, παρόλα αυτά υπάρχει φτώχεια, ε, κοινωνικός αποκλεισμός, ανεργία. Είναι λοιπόν και θέμα ευρωπαϊκών επενδύσεων. Αναρωτιέμαι εάν έχουμε εξετάσει την αποτελεσματικότητα. Ε, πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων. Είναι σημαντικό να δίδονται πόροι για τις επενδύσεις. Από την άλλη όμως μιλάμε για κάποιους πολύ περιορισμένους τομείς που δεν δημιουργούν απασχόληση. οι χώρες που τώρα βγαίνουν από την κρίση δεν επωφελούνται πολύ από αυτές τις επενδύσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε λοιπόν να επιφέρουμε μια, εξέλιξη, μια θετική εξέλιξη όσον αφορά τις επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ενεργούμε πιο αποτελεσματικά και πώς μπορούμε να κερδίζουμε περισσότερα, να επεφολούμαστε από τις επενδύσεις. Η, ε, η οικονομία ε, βελτιώνεται, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τη γραφειοκρατία και την εξάλληψή της. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Γιώζεφ Έκες από την Ουγγρική Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Πολωνό συνάδελφο και η Ουγγαρία βγαίνει από την κρίση και οι τέσσερις χώρες της Συμφωνίας Βίζικρατ μπόρεσαν να ενισχύσουν την οικονομική τους θέση χάρη στη συμφωνία αυτή. Η Ουγγαρία, όπως και η Γερμανία, έχει κάνει μια τεράστια διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Από το 2005 και μετά στηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλον. Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Από την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, τι μηνύματα λαμβάνουμε. Εάν δεν τα προσέξουμε, οι χώρες αυτές πολύ γρήγορα θα μας προσπεράσουν. Και θα ήθελα τέλος να σας θυμίσω ότι θα πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν, να εξετάσουμε για παράδειγμα το σύστημα ε, διπλωμάτων ευρυστεχνίας μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά τα διπλώματα. Οι αποφάσει των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προώθηση της επιχειρηματικής ζωής και θα πρέπει να έχουμε δομές που να μας δίνουν πραγματικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ουγγαρία έχει στηρίξει πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην δεκαετία του 2000 λάβαμε πάρα πολλούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που συνέβαλε στα θετικά αποτελέσματα της Ουγγαρίας. Έτσι μπορέσαμε να μειώσουμε την ανεργία στο 9,3%, να μειώσουμε και το πληθωρισμό. που μας ε, ταλαιπωρεί τα τελευταία 50 χρόνια. Έχουμε πετύχει πρόοδο, ε, έχουν βελτιωθεί οι επενδύσεις, δεν είναι σαφή τα θετικά σημεία ακόμα, αλλά θα δούμε θετικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριος Πρόδρομος Προδρόμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με δεδομένη την ανάγκη κάποιων έκτακτων διορθωτικών προγραμμάτων και παρά τα τυχόν λάθη παραλήψεις αλλά και προβλήματα στο σχεδιασμό μιας πραγματικά πανευρωπαϊκής οικονομικής στρατηγικής θέμα μας είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η περίπτωση της χώρας μου, της Κύπρου, ήταν κάπως ιδιαίτερη. Αντίθετα με άλλες περιπτώσεις, το Eurogroup και η Τρόικα αποφάσισαν ότι στην Κύπρο δεν θα υπήρχε δανεισμός, βοήθεια για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος. Η ιδέα ήταν να μην πληρώσουν οι φορολογούμενοι ζημιές, λάθη των τραπεζών. Σωστή και λογική ιδέα. Το ζήτημα είναι όμως η εφαρμογή της. Πριν εφαρμοστεί για πρώτη φορά η αμφιλεγόμενη ιδέα δημιουργίας τραπεζικών κεφαλαίων από τα χρήματα των καταθετών, δηλαδή με κατάσχεση, κανείς δεν φαίνεται να διερεύνησε αρκετά ή να ήξερε τις συνολικές συνέπειες μιας τέτοιας πρακτικής. Ούτε η Τρόικα, ούτε φαίνεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι συνέπειες ξεπερνούν το χρηματοοικονομικό σύστημα και το τραπεζικό πεδίο. Το ζήτημα είναι οι εξωτραπεζικές συνέπειες της τραπεζικής διόρθωσης συριγνώνοντας διαμιά το κυπριακό τραπεζικό σύστημα κατά περισσότερο από 100% και εφαρμόζοντας bail in το τραπεζικό σύστημα της χώρας βρέθηκε μετέωρο και σε αναστολή. Δημιουργήθηκε μια άνευ προηγουμένου κρίση εμπιστοσύνης. Η οικονομία αντιμετωπίζει σχεδόν απόλυτη έλλειψη ρευστότητας. Η Κύπρος μια μικρή οικονομία που χρειάστηκε δανεισμό για πρόγραμμα δημοσιονομικής διόρθωσης δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ έχει βρεθεί σε κατάσταση χρηματοδοτικής ασφυξίας. Εφαρμόζοντας επιτυχώς το πρόγραμμα διόρθωσης και ξεπερνώντας μέχρι στιγμής και αυτούς τους στόχους της Τρόικας, η πραγματική οικονομία βλέπει να βαθαίνει ύφεση και να αυξάνεται ακατάσχετη η ανεργία. Δηλαδή η πραγματική οικονομία δεν μπορεί μέχρι στιγμής να επωφεληθεί από την δημοσιονομική και την τραπεζική εξυγίανση. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα χρηματοδότησης σε πλήρη ε, αντίφαση τελικά με τον πραγματικό στόχο και σκοπό του προγράμματος. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει ο κύριος Σαχινίδης από τη Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ κάποιες χώρες της Ευρωζώνης μετά το ξέσπασμα της κρίσης διαπίστωσαν ότι η ενιαία νομισματική πολιτική τελικά μπορεί να μην είναι ενιαία. Είναι πιθανό σε συνθήκες κρίσης να έχουμε νομισματική πολιτική δύο και τριών ταχυτήτων. Έτσι, η χαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθόλου δεν βοηθά τις χώρες σε πρόγραμμα όπου οι επιχειρήσεις δανείζονται με πολύ υψηλά επιτόκια της τάξης του 8 με 10% όταν επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές χώρες δανείζονται με 4 έως 6%. Σήμερα, παρά την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και καλύπτουν το έλλειμμα ρευστότητάς τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν πάρει από το ευρωσύστημα περισσότερο από 70 δισεκατομμύρια αλλά το ευρωσύστημα πιέζει τις ελληνικές τράπεζες να επιστρέψουν πίσω το μεγαλύτερο μέρος από αυτήν τη ρευστότητα. Άρα, για όσο διάστημα δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές, δεν θα μπορούν να δανείζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για μια ανάπτυξη χωρίς πιστώσεις, ο αγγλοσαξονικός όρος είναι το creditless recovery, πόσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό το ενδεχόμενο σε χώρες σε πρόγραμμα όπως είναι η Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ε, δίνουμε το λόγο στον κύριο Σικλούνα για να απαντήσει στον πρώτο κύκλο των ομιλητών και επανερχόμαστε με τους υπολείπους. Κύριε Σικλούνα, έχετε το λόγο. Well, most of them were comments and... Uh, Τα περισσότερα σχόλια ήταν βέβαια και αυτό που είναι πολύ ωραίο στη συζήτηση αυτή είναι ότι τώρα περνάμε από το παρελθόν στο μέλλον. Πριν δούμε τη ζημιά που προκάλεσαν κάποια προγράμματα, κοινωνική ζημιά, δηλαδή ανεργία, μείωση επενδύσεων, ζημιά στο ΑΕΠ, μπορούμε να δούμε πώς θα επιδιορθώσουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε βέβαια να τα βάλουμε όλα σε ένα σακούλι. Καταρχήν πρέπει να δούμε τις μεγάλες εταιρείες που επηρεάζονται από την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να ισχύει. Ε, παίρνουν χρηματοδότηση από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και οι τράπεζες από την άλλη δεν διοχετεύουν τα κονδύλια που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το θέμα που μόλις τώρα ακούσαμε. Και μετά βλέπουμε πολλά εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη που είναι έτοιμες να επενδύσουν γιατί έχουν μικρές αγορές τις οποίες πιστεύουν και μπορούν να κρίνουν και να αναλάβουν το ρίσκο αλλά μετά ε, στερεύουν από λεφτά και εκεί παίζει ρόλο η Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι σημαντικό όμως να στοχεύσουμε την παραγωγική επένδυση. Θυμάμαι όταν ήμουν στην, Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή ε, δεν ε, ε, μιλούσαμε για τις επενδύσεις ούτε στο six-pack το πακέτο των έξι νομοθετημάτων όπου έμπαινε, έβγαινε, διαγραφόταν. Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούσαν ο, τότε ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες όταν μειώνουμε τις δαπάνες. Υπάρχουν όμως δαπάνες και δαπάνες, όπως υπάρχουν και επενδύσεις και επενδύσεις. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ τρέχει ακόμα το μνημόνιο και υπάρχουν μειώσεις στις κρατικές δαπάνες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί θύλακοι ευκαιριών όπου οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες και οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να στοχεύσουν. Διότι εδώ πρόκειται για το μέλλον μας, για παραγωγικές επενδύσεις. Αν δεν τα κάνουμε αυτά θα παραμείνουμε ε, σε υψηλή, καθεστώς υψηλής ανεργίας για περισσότερα χρόνια. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των μιλητών. Η κυρία Μπάρμπαρα Λέτσι από την Ιταλική Γερουσία, παρακαλώ. Σίγουρα επικροτούμε τις νέες επενδύσεις που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα θέλαμε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρώπη να παρέμβει με πιο μαζικό τρόπο στον έλεγχο των κυβερνήσεων και των τραπεζών. Διότι εδώ διαπίστωσα ότι μιλούν πολλές Ευρώπες. Εγώ μπορώ να συνεισφέρω το μικρό μου λιθαράκι από την εμπειρία της Ιταλίας. Ε, για πολλωστή φορία ε, κατακαιρματίστηκαν οι πιστώσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ο θεμελιώδης ιστός της ε, Ιταλικής οικονομίας και αυτή τη στιγμή έχουν γονατίσει και λόγω ε, ε, προβλημάτων που φτάνουν στο 70% της μείωσης της χρηματοδότησης. Έχουμε ένα κράτος το οποίο αυξάνει συνεχώς το δημόσιο χρέος, αυξάνει συνεχώς ε, τις μη παραγωγικές δαπάνες και μειώνει τις δαπάνες για τις επενδύσεις. Ελοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος όταν θα γίνουν αυτές οι συμπράξεις να βρεθούμε και έξω από αυτή τη βοήθεια η οποία θα βοηθήσει για τις διαθροτικές ε, μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πέραν του νομοθετικού πλαισίου στο οποίο θα μπορούσαν να κάνουν προσλήψεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας αν δεν έχουν μια αγορά στην οποία να δραστηριοποιηθούν ελάχιστες δυνατότητες θα έχουν να προσλάβουν νέους ανθρώπους διότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία είναι ότι επιχειρήσεις μας, οι οποίες ε, κατά τα δύο τρίτα θα έπρεπε να μπορούν να υποστηρίζονται από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αν δεν μπορούν να ε, χρηματοδοτηθούν, ε, θα τους επιβάλλουμε και επιπλέον όρους. Κάτι το οποίο δεν κάνουμε με τις τράπεζες. Με τη Νέα Βασιλεία υπάρχουν ε, δυνατότητες... να υπάρχει ένα 3% σε σχέση με το κεφάλαιο και, το ενεργό, και τα αποθεματικά τους. Αυτά τα εκμεταλλεύονται οι μέτοχοι των τραπεζών. Ζητώ λοιπόν μία πιο ισχυρή παρέμβαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να διασώσουν αυτή τη στιγμή την πραγματική οικονομία της Ιταλίας η οποία ε, ενώπιον μια κυβέρνηση που κάνει ελάχιστα και που διευκολύνεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία κοφεύει ενώπιον ε, των ε, προβλημάτων. Δόθηκε και ένα δις πρόσφατα για ad hoc για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε ελάχιστες εκλογικέ ομάδες. Υπάρχει μία αθέμητη πρακτική ενώπιον των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες ε, πρέπει να κατεπηγόντως να χρηματοδοθούν για να πληρώσουν το 1 τρίτο αυτών που τους οφείλεται. Η, κυβερ κυβέρνηση και το κοινοβούλιο ακόμα δεν γνωρίζει ποια είναι η πραγματική χρηματοδότηση που δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναφέρεται στην Ευρώπη και ε, δεν κάνει τα όσα θα έπρεπε να κάνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την άποψή μας. Ε, το λόγο έχει ο ε, Ογκουστέν από την Πολωνική Γερουσία. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι σε αυτή τη συζήτηση. Να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το οικονομικό και το κοινωνικό μοντέλο αποτελούν πρότυπο για πολλά μέρη του κόσμου. Και στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που διαμαρτύρονται στον Κίεβο. αποτελούν πρότυπο για πολλές χώρες. Πολλοί ακολουθούν το παράδειγμά μας. Άλλωστε έχουμε υψηλό βιωτικό επίπεδο. Δεν χαρακτηρίζει λοιπόν μόνο η κρίση την Ευρώπη. Θα πρέπει να σκεφτούμε το συνολικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι υπάρχει μια έλλειψη στη σημερινή μας συζήτηση. Εάν κοιτάξουμε τις ε, χρηματοοικονομικές αγορές, ε, θα δούμε ότι υπήρξαν κάποια, κάποιοι παράγοντες ε, που επιδίνωσαν την κρίση, αλλά και η παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει τις αγορές. Έχουμε προβλήματα με τις τράπεζες, έλλειψη εμπιστοσύνης. Και επίσης είμαστε ευάλωτοι με πολλούς τρόπους. Δεν είμαστε μόνοι μας όμως, μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να δημιουργήσουμε βιώσιμη μακροοικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε μαζί. Επίσης, έχουμε την δημογραφική ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο μπορεί να προωθήσει ή να εμποδίσει την ανάπτυξη. Και η παροχή ενέργειας σε λογικές τιμές είναι κάτι που καθυστερεί την οικονομική ανάπτυξη. Εάν δεν ενεργήσουμε γρήγορα, τότε θα επιδεινωθεί η ανάπτυξη και μπορεί να έχουμε πάλι ύφεση. Η Πολωνία συνεχώς προσπαθεί να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών. Θα ήθελα επίσης να πω ότι από τη συζήτηση αυτή προκύπτει ότι υπάρχουν προβλήματα στις κοινωνίες που δεν θέλουν να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. Και ρωτώ, υπάρχει εδώ κάποιο είδους σύγκρουση. Πρέπει να γίνουν τόσο σημαντικές περικοπές στην πρόνοια ή μήπως μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το μοντέλο αυτό. θέλουμε περικοπές. Φυσικά πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης προγράμματα υποστήριξης των νέων ανέργων. Αυτά είναι πολύ θετικά. Ε, θα κλείσω λέγοντας ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη γενικά. Διότι αλλιώς θα δούμε κοινωνικές εντάσεις, κάτι πρέπει να αποφύγουμε. Από την Ιταλική Yes, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, αν δούμε τα προηγούμενα χρόνια, αφορά τις επενδυτικές τάσεις. Αν δούμε το 2008, τότε που άρχισε η κρίση, το επίπεδο των επενδύσεων στη ΣΥΠΑ είναι ψηλότερο από το αντίστοιχο στην Ευρώπη. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε εκείνο το επίπεδο. Όταν μιλάμε για πραγματική οικονομία λοιπόν, παίζει ρόλο το πώς θα κάνουμε τις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Αυτό είναι προτεραιότητα, γιατί ε, είναι μέτρο προσφοράς και ζήτησης, ταυτόχρονα που μπορεί να ωφελήσει πολύ ε, την οικονομική ανάκαμψη. Ξέρουμε ότι οι επενδύσεις ήταν στην καρδιά του Συμφώνου Ανάπτυξης τον Ιούνιο του 2012. Πάνω από 120 δις ευρώ είχαν υποσχεθεί από το σύμφωνο εκείνο για να δοθεί ε, όθηση στις επενδύσεις. Όμως ε, το σύμφωνο ανάπτυξης είναι στα χαρτιά ακόμα. Σίγουρα αυτά που κάνει η τραπεζά σας είναι σημαντικά, αλλά δεν αρκούν. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσετε στην πρόθεση των επενδύσεων και δεν ξέρω γιατί δεν συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρόταση να υπάρξουν ομόλογα δεσμευμένα σε προγράμματα που θα τα εγγυάται η τράπεζα και θα σκοπεύουν στην υλοποίηση υπερεθνικών δικτύων, διασυνοριακών προγραμμάτων θα μπορούσε έτσι να υπάρξει κινητοποίηση πολύ περισσότερων πόρων από εκείνους που επιτυγχάνουν τα πιλωτικά προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που παρουσιάστηκαν παλιότερα. Αυτό προσκουρεί στην αντίθεση κάποιων κρατών μελών, το ξέρω, ιδιαίτερα αυτοί που δίνουν τα χρήματα. Αλλά καλό θα ήταν να γίνει με προσπάθεια τουλάχιστον να ξαναμπεί στο τραπέζι αυτή η πρόταση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη. Δεύτερον, πάλι μιλώντας για τις επενδύσεις. Πριν από λίγο καιρό, ο πρόεδρος Μπαρόζο μίλησε για ε, ένα μήνυ χρυσό κανόνα, δηλαδή να μην συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό ή δαπάνες συγχρηματοδότησης προγραμμάτων στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής κατασκευή ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Να λοιπόν μια πολύ χρήσιμη ευελιξία που θα ωφελήσει το εθνικό επίπεδο. Α, τόσο ο μήνυ χρυσός κανόνας δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα. Και όπου χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε με υπερβολικούς περιορισμούς άλλου τύπου. Η πρόταση αυτή θα μπορούσε επίσης να συζητηθεί λοιπόν για την προώθηση των επενδύσεων. Πολύ. Ε, το λόγο έχει από το Βελγικό Κοινοβούλιο ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εδώ στο Βέλγιο διαπιστώνουμε ότι έχουμε μείωση των επενδύσεων και επιβράδυνση της οικονομίας. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να δούμε και τα αίτια πέραν της κρίσης του 2008. Υπάρχουν και κάτι το οποίο δεν έχουμε αναφέρει η πολιτική της λιτότητας, ε, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μόνο ε, μέσω της αναζήτησης νέων εσόδων και επίσης ε, το γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν διαδραματίσει το ρόλο της χρηματοδότησης της οικονομίας έκαναν πιο επικίνδυνες τοποθετήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, κάτι το οποίο οδήγησε στην κρίση του 2008. Και φυσικά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μηνθούμε σε αυτά τα φαινόμενα. Αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ε, των δημόσιων μέσεων. Ε, η Τραπεζική Ένωση ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, πόρο απέχουμε και θα πρέπει ε, οι τράπεζες, λέγεται, να αποφύγουν την ιστορική τους αποστολή, δηλαδή τη χρηματοδότηση ε, σε επιχειρήσεις και σε ανθρώπους. Και υπάρχουμε, αφήνουμε, αφήνουμε από εκεί και πέρα να κερδοσκοπούν οι αγορές ε, και να μην ε, κάνουμε πραγματική χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Αναφερόμαστε συνέχεια στην πρόληψη και να προηγούμε την πρόληψη της επόμενης κρίσης και θα πρέπει οι τράπεζες να διαδραματίσουν εδώ το σημαντικό τους ρόλο, την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επίσης να δημιουργήσουν δημιουργήσουμε το κατάλληλο πρόέσιο για τη δημιουργία επενδύσεων. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις κοινωνικές πτυχές. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να μπορούμε να προασπίσουμε το οικονομικό μας μοντέλο μέσω της δημιουργίας κατάλληλων κοινωνικών δικαιωμάτων και ε, να προσπαθήσουμε να έχουμε και περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες ε, καλύτερες για τρίτες χώρες οι οποίες εισάγουν προϊόντα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν την παραγωγή προς όφελος των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε λοιπόν και κάποιους ποιοτικού δείκτες. Ε, ε, αυτή είναι και μια τεράστια πρόκληση και για το περιβάλλον και για το κλίμα. Στο Βέλγιο κάθε χρόνο έχουμε 20 δις ε, για πετρέλαιο, άνθρακα, θέρμανση μέσα αυτών των πηγών. Αν καταφέρουμε λοιπόν να έχουμε καλύτερη δυνατότητα θέρμανσης των σπιτιών μας μέσω άλλων μέσων, μέσω χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν θα χρειάζεται να επενδύσουμε αυτά τα 20 δις ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορέσουμε ίσως να βελτιώσουμε την οικονομία μας και να έχουμε καλύτερα πράγματα για το ευρωπαϊκό όραμα. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Καριμάκη από τη Φιλανδική Βουλή. Arvoisa Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σχετικά με την πράσινη οικονομία στις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τι κάνετε για τις νέες πηγές ενέργειας και την απόδοση της ενέργειας στις επενδύσεις. Αυτά οδηγούν σε ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας που οδηγεί σε αύξηση της, των εξαγωγών, θέσεις απασχόλησης ε, και ταυτόχρονα καταπολέμηση της ε, αλλαγής του κλίματος. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στο μέλλον του ευρώ και τα σχετικά μέτρα. Πολλές παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την λογοδοσία και την απόδοση ευθυνών. Ξέρουμε ότι πολλά προβλήματα οφείλονται στην υπερβολική κατανάλωση ε, και τα καταναλωτικά δάνεια. Η Φιλανδία έχει αναλάβει μέρος της χρηματοδότησης ε, του μηχανισμού για την ε, καταπολέμηση της κρίσης ε, θα ήθελα να ρωτήσω όμως ε, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε το μέλλον ε, του ευρώ. Δεν είναι απλή η απόφαση αυτή. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας για τους πολίτες, αλλά και στη Φιλανδία ακόμα έχουμε φτώχεια, ανεργία των νέων, ανεργία διαρκείας κλπ. Μειώνεται η, συγγνώμη, η φιλανδική κυβέρνηση μόλις ε, έχει λάβει απόφαση για ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων ε, που θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα στις επόμενες ε, χρονιές. Θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει το μέρος της ευθύνης του αναλαμβάνοντας μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καριέλο από την ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα σήμερα να επισημάνω ότι γίνεται αναφορά σε μία μέθοδο του μαστιγίου και του καρότου, που είναι μία μέθοδος που εφαρμόζουμε σε ζώα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν να τους μετεχειριζόμαστε σαν ζώα. Αναφέρομαι στη ρήτρα για τις επενδύσεις, βάσει της οποίας στην ε, συνεδρίαση της 22ης ε, Νοεμβρίου του Eurogroup, αναφερόμενος στην Ιταλία ότι η πρόεδρος της Επιτροπής Όλη Ρεν επιβεβαίωσε ότι η πορεία ε, των προβλέψεων για το έλλειμμα της Ιταλίας το 2014 θα οδηγήσουν σε μια δυναμία για την Ιταλία να χρησιμοποιήσει αυτή τη ρήτρα για τις επενδύσεις. Το να λέμε λοιπόν σε μια χώρα ότι αν δεν σεβαστεί τις συμφωνίες ποινικοποιούνται οι επενδύσεις για τη χώρα σου και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις επενδύσεις, σημαίνει ότι εκβιάζουμε τη χώρα αυτή. Η Ιταλία δεν θα υποκύψει σε αυτόν τον εκβιασμό, διότι αυτό σημαίνει ότι ε, μεταχειριζόμαστε τα κράτη-μέλη σαν ζώα με τη μέθοδο του μαστίγιου και του καρότου, που είναι για να τιμωρούμε τα ζώα και να συμμορφώνονται τα ζώα. Πρέπει λίγο να μετριαστεί ο τρόπος με τον οποίο ε, γίνονται επενδύσεις μεταξύ των κρατών μελών η Ιταλία, όπως και άλλες χώρες, κάνει τεράστιες θυσίε για να μπορέσει να σεβαστεί τα όρια και είναι αντικείμενο αυτού του εκβιασμού, ο οποίος ε, εφαρμόζεται αδιακρίτω, ανεξάρτητα από την οικονομική και πολιτική κατάσταση τη χώρα στην οποία απευθύνεται. Σε αυτό λοιπόν το πρίσμα της ε, αμφίβολης νομιμοποίησης, ε, στην οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη αναθεώρηση των συμφωνιών, ώστε επίτροποι όπως ο κύριος Ρέν να μην καταχρώνται την εξουσία τους και να υπάρχει ένας κατάλληλος σχεδιασμός των επενδύσεων που είναι χρήσιμες επενδύσεις για την οικονομία των κρατών μελών και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Άντερσον από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συχνά μιλάμε για τις αιτίε ε, της κρίσης, ε, γιατί ήταν ε, τόσο έντονη η κρίση. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν τεράστια όρεξη για πιστώσεις, η οποία δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί. Η αξιοπιστία της οικονομίας της Ευρώπης χάθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, διότι ε, ζούσαμε πάνω από τις ικανότητές μας. Υπάρχουν όμως ελπίδες ότι η Ευρώπη θα αποκατασταθεί και ότι θα αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη. Όλες οι χώρες έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν, να αναπτυχθεί η οικονομία τους. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην ε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Ευρώπη δεν επιτρέπεται με την γραφειοκρατία να εμποδίσει, να αναπτυχθούν οι δυνατότητες της κάθε χώρας. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε την δυνατότητα καινοτομίας και ανάπτυξης. Οι πολίτες δημιουργούν τις θέσεις εργασίας. Πολύ λίγες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από πολιτικούς. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις για περισσότερες ελευθερίες. Ε, θα πρέπει να σώσουμε τις θέσεις εργασίας, να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα και έτσι να κινητοποιήσουμε και τις επενδύσεις. Τούτου λεχθέντος ε, θα πρέπει να δώσουμε βάρος ε, στην μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε κάθε χώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλώ τον κύριο Σικλούνα να απαντήσει στον δεύτερο κύκλο των ομιλητών πριν διακόψουμε. Um, λοιπόν, έγιναν διάφορες παρατηρήσεις. Μία αφορά τις αποτυχίες στην αγορά, δηλαδή οι τράπεζες λόγω των υπερβολικών κανονισμών που αντιμετωπίζουν, των υπερβολικών ρυθμίζεων, ε, ασχολούνται περισσότερο να περάσουν την αξιολόγηση παρά να δώσουν δάνεια. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες επενδυτικές, διδανειοδοτικές, καινοτομιών, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε, δηλαδή να δώσουμε εγγυήσεις. Και αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς της τράπεζας ε, με την προϋπόθεση ότι θα παρέμβει μεταξύ του δανειοδότη και της ΜΜΕ και θα δώσει τις εγγυήσεις για το ρίσκο που ναι μεν υπάρχουν στο χαμηλό επίπεδο αλλά δεν υπάρχουν σε ευρωπαϊκό. Δηλαδή, δεν ε, βλέπει ρίσκο η τράπεζα να παρέμβει σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, το θέμα των ομολόγων που συνδέονται με projects, με έργα. Δουλέψαμε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, ως πρώην Ευρωβουλευτής θα έλεγα ότι απογοητευτήκαμε που δεν δόθηκε μεγαλύτερη συνέχεια σε αυτό το τομέα. Ένας Ιταλός συνάδελφος είπε, μίλησε για τον ε, μήνυ χρυσού κανόνα. Αυτό στηρίζεται στην αρχή ότι παρά τις αναγκαίες περικοπές δαπανών, παρόλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς όπου δεν πρέπει να περιοριστούν οι δαπάνες. Πρέπει να προστατεύονται αυτοί οι τομείς. Και εδώ έχουμε και την ευκαιρία για επενδύσεις μην ε, το παρακάνουμε με τα μέτρα και χαλάσουμε και τα θετικά που υπάρχουν. Όμως οι κυβερνήσεις έκοψαν τις δαπάνες ε, για να ε, επιτύχουν τους στόχους. Δεν πρέπει όμως να περιορίζονται οι δαπάνες σε τομείς αναπτυξιακούς, γιατί έτσι καταδικάζεται η χώρα να έχει χαμηλή ανάπτυξη και απασχόληση. Και σταματώ εδώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, α, και κάποια συμπεράσματα. Ναι, συμπερασματικά πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Δεν αρκούν αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές της ανεργίας που ναι μεν φαίνεται να σταθεροποιήθηκε αλλά σταθεροποιήθηκε σε πολύ ψηλά, απαράδεκτα ψηλά επίπεδα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, εγώ δεν είμαι ο πρόεδρος της τράπεζας, είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ε, και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό το τομέα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Δεν μπορούμε να καθόμαστε άπραγοι. Και σε αυτό το σημείο διακόπτουμε για το ε, γεύμα, το οποίο υπενθυμίζω ότι είναι στον πρώτο όροφο. Επανερχόμαστε στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ.